Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ, γιατί έχουμε πολλούς προσκεκλημένους ε, σήμερα το πρωί. Θα ήθελα όλοι να έχουν ε, την, το χρόνο να τοποθετηθούν. Θα ευχαριστήσω την κυρία Ζωέλ Μικέ, είναι Υπουργός Απασχόλησης και Ισότητας και εκπροσωπεί την ε, Βελγική Προεδρία. Θα σας δώσω το λόγο ευθύς αμέσως, πριν όμως θα καλωσορίσω και τους διαδόχους σας. Θα έχουμε την Ουγγρική Προεδρία μετά τη Βελική Προεδρία. Και έχουμε την τιμή ε, σήμερα να έχουμε τρεις υπουργούς μαζί μας από την επερχόμενη Ουγγρική Προεδρία θα παρακολουθήσουν την συνεδρίαση στα πλαίσια της προετοιμασίας ο κύριος Μίλκος Μέντλινγκ, Υπουργός Ανθρωπίνων Πόρων, ο κύριος Μίλος Ζολτάης, Υφυπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων και ο κύριος Τσάντας Σόμπας, Υφυπουργός Απασχόλησης. Καλωσορίσατε. Ελπίζουμε να είναι χρήσιμη συνεδρία και για σας και για μας. Ας μην καθυστερώ λοιπόν. Θα δώσω το λόγο στην Υπουργό. Θα κάνουμε πρώτα μία ανταλλαγή απόψεων μαζί σας και κατόπιν με άλλα μέλη της ε, κυβέρνησης ε, του Βελγίου αρμόδια για τα ζητήματα που απασχολούν την Επιτροπή μας. Σας παρακαλούμε μην μακρηγορήσετε γιατί θα έχουν πάρα πολλές ερωτήσεις ε, τα μέλη της Επιτροπής μας στη συνέχεια. 10-15 λεπτάκια. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Euh, euh. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να ε, ε, ε, είμαι υπόδειγμα πρώτα απ' όλα για τους Ούγγρους συναδέλφους μου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, για την πρόσκλησή σας. Είσαστε από τις πλέον σημαντικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μας απασχολούν κοινά ζητήματα, στοιχεία κλειδιά, η οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω πλήρη επίγνωση της νέα εποχή διακυβέρνησης στην οποία εισερχόμεθα σε σχέση με το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας ε, και προφανώς ε, κατά γράμμα θα ακολουθήσουμε τις ε, νέες ρήτρε και τις νέες προβλέψεις για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη νέα δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχίζει η Βελγική Προεδρία σε μια στιγμή που είναι σημαντική λόγω της βαρύτητας ε, της οικονομικής κρίσης ε, που βιώνουμε. Επίσης, λαμβάνονται πολύ σημαντικές αποφάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη στρατηγική 2020 και για τους στόχους στον τομέα της απασχόλησης και για την μελλοντική έγκριση των κατευθυντηρίων γραμμών στον τομέα της απασχόλησης αλλά και για τις αποφάσεις για την διακυβέρνηση και δι' την οικονομική διακυβέρνηση. Έχουμε μια φιλοδοξία ε, ήθιστε να λέγεται ότι είναι υπέρμετρα φιλόδοξες οι προεδρίες, αλλά οι, προ... οι φιλοδοξίες μας επιτρέπουν να έχουμε θετικά αποτελέσματα, οπότε θέλουμε η απασχόληση να βρεθεί στο, ε, ε, στην καρδιά της οικονομικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, της πολιτικής 2020 ε, και της έγκρισης και της υλοποίησης των κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση. Επίσης, η πολιτική απασχόλησης και οι συναρμόδιοι για αυτή την πολιτική θα πρέπει να βρεθούν στον πυρήνα της οικονομικής διακυβέρνησης. Ε, προφανώς θα υποστηρίξουμε την στρατηγική 2020 ε, εφόσον ε, μιλάμε για την απασχόληση μετά το απαραίτητο lobbying, την απαραίτητη άσκηση πίεσης και μετά τις 7 βασικές πρωτοβουλίες όπου διαπιστώνουμε ότι είναι εγκάρσιος και πρωταρχικός ο στόχος η απασχόληση για τους νέους, για την καινοτομία, για την έρευνα, για τις κλιματικές αλλαγές, ε, βλέπουμε ότι είναι ε, εγκάρσιος ο στόχος της απασχόλησης στα πλαίσια όλων αυτών των 7 βασικών πρωτοβουλειών και στις τέσσερις κατευθυντήριες γραμμές ε, για την κοινωνική πολιτική και για την απασχόληση βλέπουμε συγκεκριμένα πέντε ε, στόχους ε, που απορρέουν από τη στρατηγική 2020. Τα αναφέρω αυτά για να καταδείξω πόσο σημαντικό είναι η απασχόληση να είναι στον πυρήνα όλων των πολιτικών. Δεν χρειαζόμαστε μία απλή ανάπτυξη, με ανάπτυξη που θα φέρει απασχόληση και που θα φέρει ποιοτικές θέσεις απασχόλησης. Και σε επίπεδο πολιτικό και σε επίπεδο διακυβέρνησης ε, ε, είναι σημαντικό να αναφερόμαστε στην απασχόληση. Et puis après, j'expliquerai quelles sont les grandes priorités en termes politiques euh, de la présidence. Η Βελγική Προεδρία λοιπόν θεωρεί ότι είναι ε, ε, απαραίτητο να ασχοληθούμε με την απασχόληση για να απέλθουμε από την κρίση, την οικονομική κρίση και για να υλοποιήσουμε τις νέες στρατηγικές στον τομέα της απασχόλησης. Επίσης, ε, θα, θα σας παρουσιάσουμε τον νομοθετικό πρόγραμμα της Βελικής και στη συνέχεια θα απαντήσω στις ερωτήσεις. Λοιπόν, ας ασχοληθούμε πρώτα απ' όλα με την οικονομική διακυβέρνηση. Προφανώς θα υπάρχουν και άλλα ζητήματα και άλλου είδου πολιτικές συζητήσεις, ε, το συνειδητοποιώ, αλλά... Είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε αυτόν τον ρυθμό, αυτή τη δυναμική που ήδη υπάρχει όλοι οι συναρμόδιοι στον τομέα της απασχόλησης, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ, ε, θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτή την πορεία. Συνήθως ήταν ο φτωχός συγγενής η απασχόληση ως προς τις υπόλοιπες πολιτικές. Τώρα θα πρέπει να ε, ε, ενισχύσουμε βάσει του άρθρου 9 και του βάση του άρθρου 148 της συνθήκης τον τομέα της απασχόλησης και για τους παρατηρητές και για τους εμπλεκόμενους φορείς, πέρα από την κοινωνική διάσταση της, ε, που φυσικά έχει ύψιστη προτεραιότητα και αλληλεπιδράσεις με λοιπές πολιτικές, ε, η απασχόληση θα μας χρησιμεύσει ούτως ώστε να επιδιορθώσουμε τις αγορές ε, και ε, θα χρειαστεί να αναπτύξουμε περαιτέρω έναν άλλο ρόλο της απασχόλησης ε, μακροοικονομικού χαρακτήρα είναι αναγκαίο να λειτουργήσουμε προληπτικά, εξάντε, μέσα από την ε, πολιτική απασχόλησης Άρα μέσα στα πλαίσια των μακροοικονομικών οικονομικών συζητήσεων και στα πλαίσια των συζητήσεων της οικονομικής διακυβέρνησης και του κύκλου εποπτείας ε, των χρηματοπιστωτικών αγορών η απασχόληση θα είναι στοιχείο κλειδί. Για την ε, προσφορά φυσικά είναι στοιχείο κλειδί για την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα, την επένδυση στους ανθρώπινους πόρους, ε, τα προσόντα, τα επαγγελματικά προσόντα και ε, μελλοντικά μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή οικονομία αν έχουν υψηλότερα προσόντα ε, οι εργαζόμενοι και αν αξιοποιήσουμε ε, τον πλούτο της ευρωπαϊκής αγοράς, του ανθρωπίνου δυναμικού Γνωρίζουμε όλοι ε, την ε, δημογραφική ε, κατάσταση στην Ευρώπη και στην αγορά εργασίας. Αν δεν δράσουμε θα έχουμε σοβαρότατα προβλήματα στο μέλλον. Ας πάρουμε την άλλη πλευρά, την πλευρά της ζήτησης. Το κόστος εργασίας είναι σημαντικό οι μισθοδοτικές πολιτικές ε, ως προς την ε, προσφορά ως προς την ε, συμμετοχή σε σημαντικούς τομείς που θα φέρουν νέες απασχόλησης, οικολογικός τομέας και νέες τεχνολογίες ή καινοτομία. Οφείλουμε να καταπολεμήσουμε το ποσοστό ανεργίας γιατί αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερο κόστος και χαμηλότερο εισόδημα. Δημοσιονομικό πρόβλημα λοιπόν, πρόβλημα ανταγωνιστικότητας, ε, Αυτά είναι τα δεδομένα και άρα η, πολιτική απασχόλησης εγγράφεται πλήρως ε, στα πλαίσια της οικονομικής διακυβέρνησης. Στο άτυπο συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας τονίστηκε αυτό το σημείο. Είχαμε καλέσει και τον κύριο Φανερόμπη. και μας μίλησε για τις μελλοντικέ αποφάσεις για την οικονομική διακυβέρνηση για τον Οκτώβρη και τις συστάσεις ε, της ε, ομάδας σκέψης της Task Force που έχει συσταθεί. Και εδώ φυσικά συνδέουμε το θέμα της απασχόλησης με τη μακροοικονομική εποπτεία. Υπάρχουν δύο διαφορετικές προτάσεις εξάλλου από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βασιστώ όχι μόνο στο άρθρο 121 και στο άρθρο 148 της συνθήκης. Ο στόχο είναι το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ να μπορέσει να τροποποιήσει και να βελτιώσει την μακροοικονομική ανάλυση, την προετοιμασία δικτών και ε, ο απότερο στόχος είναι να εκπονήσει συστάσεις ε, και ε, το ίδιο και για το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ πριν από το Εαρινό Συμβούλιο που θα σχετίζονται φυσικά και με το πρόγραμμα σταθερότητας και όλα αυτά πριν τη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου ούτως ώστε οι συστάσεις να σχετίζονται με την απασχόληση, αυτά για το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ, πριν περάσουμε στις συγκεκριμένες συστάσεις αναχώρα. οι συστάσεις ε, δεν μπορούν να έχουν μόνο χρηματοπιστωτικό χαρακτήρα, δημοσιονομικό χαρακτήρα, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν σφαιρικότερα ε, το θέμα της απασχόλησης. Ε, πιστεύω ότι η Επιτροπή σας θα έπρεπε να εκδώσει ψήφισμα Πάντως από κοινού ε, θα προσπαθήσουμε να σημειώσουμε πρόοδο και σε επίπεδο διακυβέρνησης και να ε, καταφέρουμε να αποκαταστήσουμε την ισορροπία ανάμεσα στην οικονομία και την απασχόληση. Ε, σε συνεργασία με τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Απασχόλησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητήσαμε συγκεκριμένες προτάσεις στο Άτυπο Συμβούλιο και σήμερα ε, θα σας παρουσιάζουμε το έγγραφο της ε, Προεδρίας μας ε, που περιέχει διάφορες ιδέες, διάφορες προτάσεις που μπορούν να ληφθούν υπόψη και κατά τη διάρκεια των εργασιών της Task Force. και πρέπει να ακουστεί η φωνή της απασχόλησης πριν ληφθούν οι αποφάσεις για την οικονομική διακυβέρνηση. Αν η απασχόληση δεν είναι στην καρδιά της λήψης αποφάσεων θα έχουμε πληθώρα εγγράφων που θα αναφέρουν την απασχόληση αλλά στην πράξη δεν θα έχουμε σημαντικά αποτελέσματα. Θα ήθελα τώρα να ασχοληθώ με τις μακροπρόθεσμες προτεραιότητες ε, της Βελγικής Προεδρίας. Βράχει πρόθεσμα έχουμε το θέμα της συζήτησης για την έξοδο από την κρίση, ε, της στήριξης, της απασχόλησης, τα μέτρα που έχουν λάβει πάρα πολλά κράτη-μέλη για την αύξηση θέσεων απασχόλησης. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε έναν ισορροπημένο διάλογο για να αποκατασταθεί η ισορροπία στην αγορά εργασίας. Ε, δεν πρέπει να δράσουμε πρόωρα γιατί είναι ακόμα αδύναμες οι αγορές ε, ίσως ε, έχουμε εμπλακεί σε αυτή τη λογική της λιτότητας ε, που είναι υπερβολική. θα ήταν πρόωρο λοιπόν ίσως να αναλάβουμε τώρα μέτρα κατά της κρίσης. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει παρακολούθηση υλοποίηση τέτοιων μέτρων και θα προκύψει και σχετική έκθεση που θα συζητηθεί στο Συμβούλιο των Υπουργών Απασχόλησης την 21η Οκτωβρίου. Θα μιλήσουμε για την περίοδο μετά την κρίση, για, τις, για τα επόμενα 5 και 10 χρόνια και τις προοπτικές για την απασχόληση, αλλά ακόμη έχουμε 23 εκατομμύρια ανέργους και θα φτάσουμε το 10% σε ποσοστό ανεργίας στην Ευρώπη παρά είναι δίνει η θέση στην οποία βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην ασχοληθούμε και με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα. Λοιπόν, τώρα για τα μακροπρόθεσμα μέτρα. Για την έξοδο από την κρίση θα χρησιμοποιήσουμε τις κατευθυντήρες γραμμές για την απασχόληση, θα σχολιάσω και την έγκρισή τους. Επιθυμούμε να προετοιμάσουμε τους, το σημαντικό διάλογο για τις διαρθρωτικές αλλαγές, που σχετίζονται με την ε, αύξηση του προσδόκιμου ζωής ε, και ταυτόχρονα την ε, μείωση της προσφοράς θέσεων απασχόλησης. Τον Οκτώβρη θα, το Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τις κατευθυντήριες γραμμές της απασχόλησης. Ο κύριος Γιούρη έχει ήδη συναντηθεί με εκπροσώπους της Βελγικής Προεδρίας και έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα δυσαρεστήθηκαν κάποιοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί ενώ δεν έχει εκδοθεί το ψήφισμα ακόμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχουν εγκριθεί κάποιες συστάσεις στο άτυπο Συμβούλιο. Προτείνω λοιπόν να συναντηθώ αύριο, ε, ε, από αύριο όποια στιγμή θέλετε να συναντηθώ λοιπόν με τον εισηγητή για να προετοιμάσουμε τον διάλογο και να προετοιμάσουμε τις καθηγητήριες γραμμές που θα εγκριθούν λαμβάνοντας υπόψη τα, τις προτεραιότητες που προβάλλατε, τις πράσινες θέσεις απασχόλησης, παραδείγματο χάρη, τους δείκτες ή τους υποδείκτες ή τους υποστόχους. Αυτή την ορολογία χρησιμοποιούμε. Πέρα από την έγκριση των κατευθυντηρίων γραμμών, θέλουμε να προετοιμάσουμε και τις μεγάλες στρατηγικές αλλαγές στον τομέα της απασχόλησης και της οικονομικής ε, πολιτικής. Πρασινοποίηση, όπως λέμε, της οικονομίας ε, και ε, προσαρμογή του χρόνου εργασίας. Θέλουμε να προαγάγουμε θέσεις απασχόλησης με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα επιθυμούμε να προσαρμόσουμε τις θέσεις απασχόλησης ακολουθώντας αυτή τη γραμμή. Σας παραπέμπω και στο άτυπο συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας η υπουργική μας διάσκεψη που θα λάβει η χώρα στα τέλη Σεπτεμβρίου, 28 και 29 Σεπτεμβρίου, Εξάλλου θα ε, παρευρεθεί και η κυρία Σρέντερ που εκπώνησε την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεσή της για τη μετάβαση προς τις πράσινες θέσεις απασχόλησης, ε, προς την πιο πράσινη οικονομία. Θα λάβουμε και την έκθεση ΕΜΚΟ το φθινόπωρο η φιλοδοξία μας ε, σε σχέση και με τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε σχέση με τη διυπουργική διάσκεψη και του εγγράφου εργασίας, ε, του ιστορικού εγγράφου εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φιλοδοξούμε να, έχουμε, να καταλήξουμε σε φιλόδοξα συμπεράσματα ταχύτατα σε σχέση με τη μελλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την παράταση του του εργάσιμου χρόνου δεύτερη μεγάλη προτεραιότητα της Βελικής Προεδρίας. Θα διοργανώσουμε μια μεγάλη διάσκεψη ε, σε συνεργασία με το Ίδρυμα του Δουβλίνου για, τη, για αυτή την προβληματική, δηλαδή παράταση της επαγγελματική σταδιοδρομίας και ποιες συνέπειες έχει αυτό για τη, ως προς την ποιότητα της εργασίας, ε, του, της οργάνωσης της σταδιοδρομίας και ξαναλέω της ποιότητας ε, της απασχόλησης. 16 και 17 Οκτωβρίου θα λάβει η χώρα αυτή η διάσκεψη και ένα άλλο σεμινάριο για μια εξίσου σημαντική διάσταση, δηλαδή να δημιουργήσουμε ε, λευκές θέσεις απασχόλησης όπως ονομάζονται πέρα από τις πράσινες θέσεις απασχόλησης να λειτουργήσουμε προληπτικά και να κατοχυρώσουμε τις υπηρεσίες προς τους ανθρώπους και να ε, δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση λαμβάνοντα υπόψη την νέα πραγματικότητα, την παράταση του εργάσιμου χρόνου τη επαγγελματική σταδιοδρομία. Για την αναδιάρθρωση, ε, μην ξεχνάμε ότι υπήρξαν φόρες στα 27 κράτη-μέλη και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΕ στις 18 και 19 Νοεμβρίου θα γίνει ένα σεμινάριο. Ουσιαστικά πρόκειται για διάσκεψη όπου θα συζητήσουμε αυτό το θέμα και θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Δηλαδή, τι χρειαζόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να λειτουργήσουμε προληπτικά σε σχέση με τις αναδιαρθρώσεις για αυτή τη μεταβατική περίοδο προς μία αγορά εργασίας όπου οι εργαζόμενοι θα έχουν υψηλότερα προσόντα και τελειώνω ένα λεπτάκι ακόμα. Ε, πάλι για τους μακροπρόθεσμους στόχους, ε, η ευελίξη ασφάλεια, ευελιξία και ασφάλεια, η θέσει απασχόληση για του νέου, η έξοδο από την κρίση. Αναμένουμε την ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στον τομέα αυτό. και θα διοργανώσουμε μια σχετική διάσκεψη. Θα προκύψει η δήλωση της Προεδρίας και θα πάρουμε και την έκθεση της Επιτροπής σας και όλα αυτά θα συζητηθούν στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Κατά πολέμηση τη διακριτικής μεταχειρίσης στην αγορά εργασίας. Αυτό θα είναι το βασικό θέμα ε, στις 15 και 16 Νοεμβρίου που θα γίνει σύνοδος για την ισότητα των δύο φύλων. Πέρα από τις υπόλοιπες προτάσεις που θα κάνουμε για την ισότητα των δύο φύλων σε άλλα φόρα και τώρα μιλώ με την ιδιότητά μου ε, της Υπουργού Αρμόδιας για τα στήματα της ισότητας των δύο φύλων και εξάλλου θα πάω και στην Επιτροπή Γυναικών στις 11 η ώρα. Για τις νομοθετικές εργασίες ε, Νομίζω ότι ε, τώρα που θα μου θέσετε ερωτήσεις ε, θα επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, ανακεφαλαίωνο θα έχουμε τις κατευθυντήριες γραμμές. Δεύτερον, για το χρόνο εργασίας ε, δεν θα δημιου... σημειωθούν εξελίξεις κατά τη διάρκεια της Βελικής Προεδρίας γιατί προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη θέση της επί τη βάση μιας αξιολόγησης αντικτύπου της δημόσιας διαβούλευσης που γίνεται οπότε είναι μάλλον θέμα της Ουγγρικής Προεδρίας. Η μελλοντική οδηγία για την προστασία των εργαζομένων από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία με ε, μία έκθεση που περιμένουμε για τέλη Οκτωβρίου 2010 ε, και σε συνεργασία με την Επιτροπή των Γυναικών θα δούμε και την εξέλιξη της οδηγίας ε, για την άδεια μητρότητας. Ε, και επίσης ε, για την οδηγία για τη διακριτική μεταχείριση και ξέρω ότι δραστηριοποιείται και η Επιτροπή σας όλος ιδιαίτερος ε, μέσω του εισηγητή σας για τα ψηφίσματα που θα προκύψουν και για την μετανάστευση. Τώρα αλλάζω πάλι καπέλο, αλλάζω ιδιότητα. και προφανώς ε, θα κληροδοτήσουμε όλα αυτά τα θέματα στην Ουγγρική Προεδρία, ό,τι σχετίζεται δηλαδή με την προστασία των εργαζομένων μετακινούντες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαχειριστούμε αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα. Ε, καταλαβαίνετε ότι είναι περίπλοκη κατάσταση στο Βέλγιο. Έχουμε ε, σε σημαντικά προβλήματα διότι ακόμη ε, δεν ε, έχουμε κυβέρνηση. Ελπίζω ότι δεν θα καθυστερήσει αυτό. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχαμε συζητήσει μαζί σας ήδη όταν ήρθαμε να σας επισκεφθούμε, μια, ένα κλιμάκιο της Επιτροπής μας σας επισκέφθηκε. Είναι πολύ φιλόδοξο το πρόγραμμά σας ε, όντως. Τώρα, δυστυχώς, ε, πρέπει να πω ότι έχουμε 25 λεπτά στη διάθεσή μας ε, και 8 ομιλητές. Δεν μπορείτε να υπερβείτε τα δύο λεπτά. Ο κύριος Τσαβάουρη και ο κύριος Αλισάνδρος Σέρκας. Πρώτα απ' όλα, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτήν την διαφωτιστική παρουσίαση. Στον ε, τομέα της απασχόλησης νομίζω ότι βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος εδώ στο Κοινοβούλιο σε σχέση με το πρόγραμμα της Βελγικής Προεδρίας. Στην παρουσίασή σας μας μιλήσατε για την πολιτική απασχόληση και είπατε ότι συχνά είναι ε, ο φτωχός συγγενής η απασχόληση. Δηλαδή, επιδιώκουμε να βρούμε στρατηγικές εξόδου από την κρίση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να σκεφτούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την απασχόληση για να ε, βγούμε από την κρίση. Τι πιστεύετε για τις υπόλοιπες ε, πολιτικές. Δηλαδή τι χρειάζεται ουσιαστικά για να μπει στην καρδιά κάθε πολιτική η απασχόληση. Παραδείγματος χάρη, η πολιτική που θα ακολουθηθεί για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ε, πολύ μεγάλο δυναμικό. Μπορούν να δημιουργήσουν πολλές θέσεις απασχόλησης. Δεν αναφερθήκατε στο θέμα της χρηματοδότησης. Αλλά θα ήθελα εδώ να σας θυμίσω ότι η πολιτική συνοχή μπορεί να μας ε, βοηθήσει πάρα πολύ στον τομέα της απασχόλησης. Το ξέρω ότι δεν έχουμε λεφτά. Ο κύριος Σέρκας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι ως συντονιστής της ομάδας εργασίας των σοσιαλιστών θέλω να σας διαβιβάσω την επιθυμία να έχετε μια επιτυχή προεδρία και θα ήθελα να προσφέρω και τη συνεργασία μας προς αυτόν τον στόχο. Έχω την εντύπωση ότι αυτό θα γίνει, θα είναι επιτυχής η προεδρία σας διότι το Βέλγιο και η κυβέρνηση σας ε, είναι μια μεγάλη χώρα με τεράστιες δεσμεύσεις φιλευρωπαϊκές και με μεγάλη δέσμευση επίσης ε, για την κοινωνική διάσταση και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Μπορείτε να βασίζεστε στη συνεργασία μας με ειλικρινή τρόπο και με κάθε ζήλο και ενθουσιασμό. Για κάποιες ερωτήσεις ε, και που θα είχα κάποιες. Θα ήθελα να σας δώσω την ευκαιρία να υπογραμμίσετε κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ο προσανατολισμός σας που ήδη γνωρίζαμε σε σχέση με τα όσα μας ανέφερε αναφέρθηκαν και για να ενταχθούν οι εργασίες της Task Force σε σχέση με τον πρόεδρο Φαν Ρόμποϊ και σε σχέση με το άρθρο 148 128 πρώην για την ιστορική ας το πω έτσι διάσταση ώστε η απασχόληση να περάσει από την βιβλιογραφία και τη θεωρία στην πραγματικότητα των συνθήκων και να είναι η πραγματικότητα η καθημερινή για την Ευρώπη. Μακάρι να μπορέσει να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Δύο παρατηρήσεις για το νομοθετικό τμήμα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα για το θέμα της μετανάστευσης να πω κάτι. Είμαι ε, εισηγητής ε, για το ε, θέμα της single permit και παρακολούθησα το θέμα των εργαζομένων που εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Προσπαθούμε, προσπαθήσαμε κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας να γίνει η ανάγνωση, η πρώτη ανάγνωση Έλειπε όμω ένα σημαντικό στοιχείο των προσωρινών εργαζομένων. Τώρα το έχουμε. Θα μπορούσαμε από κοινού να εργαστούμε. Θα μπορούσαν οι υπουργοί ή από πλευρά του ε, Συμβουλίου που είναι αρμόδιοι να κάνουν μια προσπάθεια για να καταλήξουμε σε μια πρώτη ανάγνωση. Έχω αποστείλει μια επιστολή για την κοινωνική διάσταση από πλευρά του Single Permit. Μπορείτε να αναλύσετε αυτή την επιστολή και τι επιθυμίε μα. Ε, και από πλευρά ε, των προσπαθειών αυτών, πέρα από τις οδηγίες, θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχει κάτι για μια οδηγία, για παράδειγμα, ώστε για τα μειοσκελετικά προβλήματα αν ε, μπορεί να γίνει κάτι και για τις ε, φυσικές σωματικές επιπτώσεις και αν θα μπορούσαμε να είχαμε και για τις άτυπες μορφές εργασίες μια επαφή. Ευχαριστώ. Πουπακής, Πουπάκη, παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας και την προσπάθεια που κάνετε. Ε, σε αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, ε, βαθιάς οικονομικής δημοσιογικής κρίσης, με κοινωνικέ διαστάσει εξάπλωση φτώχεια και κοινωνικού αποκλεισμού, βλέπουμε ότι γίνονται κάποιε προσπάθειε από τα κράτη-μέλη για να βγούμε από την ύφεση, να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, με αποτέλεσμα βέβαια ε, να μειώνονται αλόγιστα κοινωνικέ δαπάνε με δυσμενεί επιπτώσει για την κοινωνική σταθερότητα και συνοχή. Για παράδειγμα, ίσω χρειάζονται διασφάλιση εξοπλισμού διαβίωση για όλου μέσα από ενίσχυση απασχόληση και προνοιακών πολιτικών, κυρίω για νέου εργαζόμενου και ευάλωτε ομάδε, διασφάλιση επαγγελματική πορεία εργαζομένων στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων επιχειρήσεων και τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικολογική οικονομία. Θα ήθελα να σα ρωτήσω, με αφορμή την κρισιμότητα αυτού του επόμενου εξαμήνου και τι προτεραιότητε που βλέπω ότι δίνεται τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική διάσταση τη Ευρώπη, πώς προτίθεστε να διασφαλίσετε αυτή την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο μερών, των δύο τομέων. Ευχαριστώ. Euh, σας ευχαριστούμε, η κυρία Λίν. Uh, uh, ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που σα ξαναβλέπω και ευχαριστώ που ήρθατε στην Επιτροπή μα Σε τρει πολύ σύντομε ερωτήσει για νομοθετική φύσεω θέμα. Αναφερθήκατε ε, στο ότι θα ήταν χρήσιμο όσον αφορά τις 18 με 20 εβδομάδες ε, πλήρους ε, διατήρησης ε, του μισθού. Μήπως μπορείτε να τοποθετείτε από αυτού, διότι πιστεύω με την οικονομική κρίση που βιώνουμε, λόγω του ότι υπάρχουν διαφορετικές νομοθεσίες και παραδόσεις στα κρατημέλη, ίσως είναι και κατάλληλη στιγμή για να προχώρησε ένα τέτοιο μέτρο. Δεύτερον, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, στο Κοινοβούλιο έχουμε ασχοληθεί με την οδηγία περί των ε, ε, σαρωτών. Έχουμε ασχοληθεί με τους δημογράφους τομογράφους ε, και θα θέλαμε να γνωρίζουμε κατά πόσον και άλλοι θα εμπίπτουν σε αυτή την οδηγία περί δεν ξέρω ε, κατά πόσον είχατε χρόνο να ασχοληθείτε με αυτή την οδηγία. Και τέλος, όσον αφορά την οδηγία κατά των διακρίσεων. Ε, κατανοώ ότι η οδηγία αυτή έχει κολλήσει στο Συμβούλιο και εμείς ε, συνεχίζουμε να διερωτώμεθα κατά πόσον υπάρχει κάποια εξέλιξη. Βεβαίως τις περισσότερες φορές μας λένε ότι δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Εσείς ε, ως Βελγική Προεδρία πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε για να ξεμπλοκάρετε την ε, οδηγία περί διακρίσεων έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Ε, συνάδελφοι, κλείνω τον ε, κατάλογο των ομιλητών ε, και ε, ήδη έχουμε τρεις ομιλητές που έχουν εγγραφεί αλλά δεν θα έχουν το χρόνο να τοποθετηθούν. Θα τοποθετηθούν στην επόμενη συζήτηση. Ο κύριος Κώσσα. Κυρία Κώσα, θα ήθελα... Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας καλωσορίσω θερμά κυρία Υπουργέ Χαίρομαι πρέπει να πω για το γεγονός ότι ακούσαμε ότι το πρόβλημα των ατόμων με μειονεξία θα εντάσσεται στην ημερησία διάταξή σας και η Ισπανική Προεδρία το είχε θέσει σε, ως προτεραιότητα αυτό το θέμα όμως δυστυχώς δεν υπήρξαν πάρα πολλά αποτελέσματα χειροπιαστά. Όταν γίνεται εδώ λόγος για την διεύρυνση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Πώς μπορεί κανείς να πετύχει μεγαλύτερη απασχόληση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με μειονεξίες. Έχει η Βελγική Προεδρία κάποιο σχέδιο υπόψη για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Δεύτερο. Το δεύτερο είναι ότι όσον αφορά τις οικογένειες και τα προγράμματα μέσα στο πλαίσιο ενός προγράμματος φιλοοικογενειακών δράσεων. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια δημογραφική αλλαγή, μεταβολή στην Ευρώπη και θα έχουμε όλο και μεγαλύτερο αριθμό όχι μόνο περιλίκων αλλά και ατόμων με μειονεξίες, με ειδικέ ανάγκες. Τι γίνεται ακριβώς με τις κοινωνικές υπηρεσίες, την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για οικογένειες, για άτομα με ειδικέ ανάγκες. Υπάρχουν προγράμματα, θα υπάρχουν προγράμματα τα οποία προβλέπει η Βελγική Προεδρία και θέλει να υλοποιήσει, διότι τα προβλήματα των οικογενειών ακριβώ είναι σημαντικά. Θα πρέπει να τύχουν προσοχή ε, τα προβλήματα των ανθρώπων με μειονεξίες που ζουν στις οικογένειές τους. Να ληφθούν λοιπόν οι οικογένειες υπόψη. Εκεί χρειάζεται μια νομοθετική πρωτοβουλία. Και μπορεί κανείς να φανταστεί ότι και μια χάρτα ευρωπαϊκή για άτομα με ειδικέ ανάγκες θα μπορούσε να θεσπιστεί ώστε η ελευθερία κυκλοφορίας και κινητικότητα των ατόμων αυτών να βελτιωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα μπορούσε επίσης να ασκήσει την επιρροή του από πλευράς του στην κοινωνική διάσταση και στις κοινωνικές υπηρεσίες, στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Είναι σημαντικό. Η κυρία Αντελή, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Υπουργό για την παρέμβασή της. Θα θέσω δύο ζητήματα. Ε, το έτος καταπολέμησης στις στόχες ε, και η όρια εργασίας. 85 εκατομμύρια φτωχούς έχουμε σήμερα ε, και είπαμε όλη τη χρονιά, όλη τη χρονιά ακουγόταν ότι οι μισοί έχουν κάποια θέση απασχόλησης. Θέλουμε να ενεργοποιήσουμε τους ανέργους, κυρίως αυτούς που έχουν απομακρυνθεί περισσότερο από την αγορά εργασίας. Αυτό είναι από τους βασικούς στόχους της Βελικής Προεδρίας. Ε, προφανώς είναι θεμητός ο στόχος, ε, αλλά πρέπει να αναγνωρίζετε ότι η απασχόληση δεν προστατεύει πλέον τους φτωχούς. Θα έχετε το βαρύ καθήκον λοιπόν να κλείσετε το έτος καταπολέμησης της φτώχειας και της κοινωνικής αποξένωσης και θέτω το εξής ερώτημα. Η Βελγική Προεδρία θα δρομολογήσει μια πρωτοβουλία ούτως ώστε να υιοθετηθεί μια ευρω... ευρωπαϊκή οδηγία για το ελάχιστο εισόδημα. Δεύτερον, ε, σχετικά με την υποβάθμιση των όρων εργασίας. 160.000 ε, ε, θάνατοι που στο χώρο εργασίας, 60.000 περιπτώσεις καρκίνου. Vous σε σχέση με αυτά που γίνεται στο, διεθνές, ε, στο Διεθνή Οργανισμό Εργασίας ε, και την οδηγία για την έκθεση στους κινδύνους των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά σχετίζονται με την κοινωνική ασφάλιση και με την έκθεση σε άλλων ειδών ουσίας, όπως σε οι καρκινογόνες ουσίες. Ευχαριστούμε κυρία Πασκάλ Γκρινή. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την Υπουργό για την παρουσία της ε, σήμερα το πρωί. Όταν μιλάμε για την επιστροφή στην απασχόληση δεν μπορούμε να ξεχνούμε το ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο Απασχόλησης. Δεν αναφερθήκατε καθόλου σε αυτό. Τώρα προετοιμάζεται το κονδύλι για την προγραμματική περίοδο το 2014 έως 2020 υπάρχουν ανησυχίες σε σχέση με την αυτονομία του Ταμείου ως προς τα διαρθρωτικά ταμεία, την απλούστευση της διαδικασίας. Συζητώντας λοιπόν αυτό το κονδύλι θα είχατε κάτι να προσθέσετε και σε σχέση με αυτό που μας είπε η κυρία Λίν για τις 18 ως 20 εβδομάδες. Ναι, αλλά ποιο θα είναι το ποσοστό αποζημίωσης, ποιες θα είναι οι αποδοχές. Και όπως είπε και η κυρία Καρή Μαντελή, μας απασχολεί η υγεία και η ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Ε, τα δύο τρίτα των επαγγελματικών δεδηλωμένων νόσων οφείλονται σε μειοσκελετικές διαταραχές. Ε, θα είχατε κάποιο σχόλιο να κάνετε. Πρόεδρος. Δεν ε, είμαι σίγουρη ότι θα έχει χρόνο να απαντήσει όλο όλα ο υπουργό, αλλά τουλάχιστον θα έχει το χρόνο να τα ακούσει όλα. Ο κύριος Στέφεν Χιούζε και η κυρία Άρκιν. Στέφεν Χιούζε. Πρόεδρε, δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις. Πρώτον, όσον αφορά το θέμα της απασχόλησης, ε, η οποία πρέπει να είναι το κύριο μέλημα στη μακροοικονομική πολιτική. Προφανώς συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας, αλλά πώς θα μπορέσετε να πείσετε το ΕΚΟΦΗΝ ότι κάτι τέτοιο πρέπει να ισχύει γιατί αυτοί επιθυμούν να μειώσουν το έλλειμμα στο 3% για όλα τα κρατημέλη μέχρι το 2013. Οι σοσιαλδημοκράτες ε, πρότειναν να υπάρχει σε όλο αυτό το θέμα και ένα πακέτο απασχόλησης. Να πούμε ναι εντάξει, να μειωθεί το έλλειμμα στο 3% αλλά κανένα κράτος μέλος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει και την ανεργία πάνω από 5% σε αυτό το δρόμο που θα ακολουθήσει. Έχετε εσείς συγκεκριμένες προτάσεις που θα μπορούσαν να αλλάξουν ε, αυτή την ισορροπία που υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάμεσα στην απασχόληση και την ε, μείωση του ελλείμματος. Δεύτερη ερώτηση. Είστε σίγουροι ότι οι αυτοπασχολούμενοι οδηγοί συμπεριλαμβάνονται και αυτοί στο καθεστώ του ωραρίου εργασία. Εκτό αν γνωρίζω, στο Συμβουλίο υπάρχουν όλο και περισσότερε κυβερνήσει οι οποίε λένε ότι κάναμε λάθο για δεύτερη φορά και ότι οι αυτοπασχολούμενοι οδηγοί θα πρέπει να αποκλείονται από αυτήν την οδηγία. Εσεί, η Βελγική Προεδρία, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι η Κομισιόν θα κάνει το σωστό και θα αποσύρει αυτή την πρόταση τώρα που εμεί οριστικά την καταδικάσαμε κυρία Αρκίν. Σας ευχαριστώ και πρώτα απ' όλα καλώς ήρθατε προς την Βελγική Προεδρία και κάθε επιτυχία στο πρόγραμμα εργασίας. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρετε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Δύο σύντομες ερωτήσεις. Η πρώτη είναι εκείνη που ρωτήθηκε και για τη μακροοικονομική κατάσταση από πλευρά Steven Hughes. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω εγώ την ερώτηση. Συμφωνώ με, απόλυτα με αυτά που είπε ο Στίβεν Hughes. Να προσθέσω μόνο σε αυτά και σε σχέση με τις περικοπές έχουμε και περικοπές και στον ε, δημόσιο τομέα στα κράτη-μέλη και για τις ε, υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Ίσως αυτό θα μπορούσατε να το εντάξετε στην απάντησή σας. Δεύτερη ερώτηση. Σε σχέση με την τεκμηρίωση λέγεται ότι η Βελγική Προεδρία θέλει να εξετάσει τις δυνατότητες εξέβρεσης ενός κοινού πλαισίου για ένα ελάχιστο πρόγραμμα που θα έχει ελάχιστα κριτήρια για την ε, προσπελασιμότητα και την ε, αποδοτικότητα. Μπορείτε να τα επεξηγήσετε αυτά κάπως. Ευχαριστώ κύριο Φάμπερ. Ευχαριστούμε ο κύριος Φάμπρ και η κυρία Μιζότος στη συνέχεια. Σα ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση προς την κυρία Υπουργό, αν επιτρέπετε. Και αυτή αφορά μια οργάνωση που είναι ξεχωριστή. Μια βελγική ε, οργάνωση που θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη, θα έχει επίπτωση αυτός ο σύλλογος, αυτή η ένωση και πώς έχετε υπόψη να συνεργαστείτε μαζί τους και με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Merci, Madame Bizotto. Ευχαριστούμε κυρία Μιζωτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ο στόχος σας είναι να ενισχύσετε περισσότερο το κοινωνικό μοντέλο. Όμως ε, δεν είναι ουσιαστικά σημαντικότερο να ε, ε, θέλετε να τροποποιήσετε το κοινωνικό μοντέλο. Παραδείγματο χάρη στο Βέλγιο υπάρχει ένα πολύ γενναιόδωρο κοινωνικό κράτος που προβλέπει και πάρα πολλά επιδόματα για τους ανέργους. Αυτό δηλαδή το μοντέλο προτίθεστε να προτείνετε και τι πιστεύετε για το ελάχιστο κειμένο ισότητα και μια άλλη ερώτηση που αφορά στι μειονότητε και στα δικαιώματα των γυναικών. Εγώ έκανα μια ερώτηση στην Κομισιόν όσον αφορά το θέμα τη Μπούρκα. Και μου απήντησαν ότι μεταξύ άλλων ε, σαφώς και πρόκειται για παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών. Εμείς γνωρίζουμε ότι το Βέλγιο όπως και η Ισπανία και η Γαλλία έχουν εκπονήσει τη σχετική νομοθεσία που κατ' ουσίαν απαγορεύει την Μπούρκα θα ήθελα να γνωρίζω κατά πόσο η Βελική Προεδρία σκοπεύει σε κοινοτικό πλέον επίπεδο να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την απαγόρευση της Μπούρκα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι αυτό το θέμα έχει να κάνει τόσο με την ένταξη της γυναίκας στην κοινωνία, όσο και με την ασφάλεια. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη από τρεις συναδέλφους που έχω. Είχαν ζητήσει το λόγο, αλλά ε, δυστυχώς δεν μπορώ να τους το δώσω τώρα. Θα τοποθετηθούν στην επόμενη συζήτηση. Υπουργέ, ε, έχετε λίγο χρόνο για να απαντήσετε σε αυτές τις δέκα ερωτήσεις. Είμαι σίγουρη ότι θα τα απεξέλθετε στην πρόκληση. Υπουργός, ε, κυρία Μιλκέ, ε, δυστυχώς δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Θα βάλω τα δυνατά μου. Ε, θα απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Ορή. Πρώτα απ' όλα, είναι προφανές ότι είναι εγκάρσιος ο στόχος υποστήριξης απασχόλησης και υπάρχει υποστήριξη από άλλες πολιτικές ε, όπως η πολιτική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ε, ο βασικός πάροχος δέσεων απασχόλησης αν θέλετε στην αγορά εργασίας και μέσα στην ομοθεσία της Small Business Act για τις μικρές επιχειρήσεις και στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 ε, προβλέπεται επίτευξη αυτού του στόχου, δεν είναι θέμα δικής μου αρμοδιότητας. Οι συνάδελφοί μου αναλαμβάνουν διάφορες πρωτοβουλίες ε, για να υποστηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να ε, προαγάγουν το πνεύμα της επιχειρηματικότητας. Ε, θα επανέλθω σε αυτό το θέμα και σε σχέση με ερωτήσεις που έθεσαν οι συνάδελφοί σας, αλλά πάντως όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε αμέριστη ευθύνη στον τομέα αυτό και από δημοσιονομικής πλευράς και από πλευράς επενδύσεων σε πολιτικές κλειδί κλειδιά σε επενδύσεις ε, για την ε, αύξηση των επαγγελματικών προσόντων ή ε, πολιτικές στήριξης της αγοράς εργασίας μέσα από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κύριε Σέρκας, θα συναντηθούμε για να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να εντάξουμε τις τροπολογίες σας στο εγγραφό μας και πώς θα, το, θα τη συνδυάσουμε με το, την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών ε, σε σχέση με την οδηγία για την ενιαία εργασία, το Single Permit. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό ε, για την, παράνομη, για την καταπολέμηση της παράνομης εργασίας. Επίσης, ε, σε μελλοντικές ε, νομοθετικές, ε, νομοπαρασκευαστικές συζητήσεις για την απόσπαση των εργαζομένων, ένα θέμα που θα μας απασχολεί στο 2011, οι συζητήσεις που γίνονται για τους εποχιακούς εργαζομένους, για την κοινωνική τους ασφάλιση. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις νομοθετικού χαρακτήρα που συνδέονται και με άλλα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν στην αγορά εργασίας η κατάργηση της διακριτικής μεταχείρισης, το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης, όλα αυτά τα ζητήματα είναι αλληλένδετα. Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να ικανοποιήσω τις προσδοκίες σας σε σχέση με όλες αυτές τις οδηγίες που προανέφερα τώρα. Ε, με ποιο τρόπο ε, μπορούμε να κατοχυρώσουμε μια επαρκή στήριξη στις ομάδες στόχους στα πλαίσια της πολιτικής απασχόλησης, ε, μιλώντας για τα πιο ηλικιωμένα άτομα, για την μετάβαση στην ε, οικονομία με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα, πιο πράσινη οικονομία, αλλά με υψηλότερα προσόντα. Ναι, κοιτάξτε, ε, θα πρέπει να ασχοληθούμε με τις ομάδες στόχους και με την εξέλιξη αλλαγματική πορεία της οικονομίας μας ε, θα χρειάζονται όλο ένα και υψηλότερα επαγγελματικά προσόντα. Αυτό είναι αναμφισβήτως. Σε σχέση με αυτά που μας είπε η κυρία Λίνε, η οδηγία για την άδεια μητρότητας ε, είναι λεπτό το ζήτημα, είναι ακαθόδης γιατί διαπιστώνουμε μία διάσταση απόψεων ανάμεσα στην τοποθέτηση της Επιτροπής ε, Απασχόλησης και της Επιτροπής Γυναικών, στην οποία θα μεταβώ τώρα. Μόλις ολοκληρώσα την παρέμβασή μου και αυτό σχετίζεται με θέματα προϋπολογισμού. Έχουμε πάρα πολύ σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε ε, και αν θέλετε την προσωπική μου άποψη είναι πιο λογική η προσέγγιση της Επιτροπής Απασχόλησης σε σχέση με την προσέγγιση της Επιτροπής Γυναικών. Ε, προφανώς θα συνεχίσουμε το διάλογο και με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προωθήσουμε αυτή την οδηγία. Από πλευράς μας έχουμε και εμείς κάποιες νέες ιδέες. Ε, υπάρχει και το θέμα της ημερομηνίας ε, εφαρμογής αυτής της οδηγίας που θα μπορούσε να επηρεάσει την δημοσιονομική διάσταση του προβλήματος. Πάντως στη συζήτηση θα ληφθούν ναι, ε, υπόψη οι τροπολογίες επιτροπή απασχόληση. Κύριε Πόζα, ε, μιλήσατε για τα άτομα με αναπηρίες. Ε, πολύ σωστά. Στην διάσκεψη που θα κάνουμε για την ισότητα και θα προετοιμάσουμε και συμπεράσματα που σας είπα στην αρχική μου παρέμβαση, θα ληφθούν υπόψη τα σχόλιά σας και επανέρχομαι σε κάτι που μας είπε και η κυρία Λίν. Θα θέλαμε ε, η οδηγία για τη διακριτική μεταχείριση να προχωρήσει. Επίσης είναι περίπλοκο το ζήτημα για γνωστούς λόγους. Ο στόχος είναι να επιτύχουμε ταχύτατα συνένεση μέσω μιας θεματικής προσέγγισης. Ένα από τα θέματα λοιπόν αυτής της προσέγγισης είναι ακριβώς οι αναπηρίες. Εξάλλου υπάρχει και η οδηγία για την προστασία των εργαζομένων από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Τώρα προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχετικό της έγγραφο, θα της δείξουμε εμπιστοσύνη και όταν παρουσιαστεί το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, τότε θα επανέλθουμε για να σχολιάσουμε όλα τα τεχνικά επιμέρους ζητήματα που θίξατε. Νομίζω ότι ακόμη και αν απευθυνθείτε τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορέσει να σα απαντήσει γιατί δεν έχει ακόμη εκπονήσει τη μελέτη της. Για τις αναπηρίες ε, συνιστά προτεραιότητα για μας ε, και γιατί να μην, ε, όπως σωστά προτείνατε, να μην επιδιώξουμε και μια ευρωπαϊκή χάρτα για τα άτομα με αναπηρίες. Ως προς την ε, καταπολέμηση τώρα της ε, φτώχειας και της κοινωνικής αποξένωσης θα έρθει τώρα η συνάδελφός μου, η κυρία Λορέτ Άγκελινγκς ε, που είναι άμεσα αρμόδια για τα θέματα φτώχειας. Η φτώχεια φυσικά δεν είναι ένα μεμονωμένο θέμα συνδέεται με όλες τις, ε, τις υπόλοιπες προκλήσεις ε, και θα σας μιλήσει η συνάδελφός μου για το θέμα του ελαχίστου εισοδήματος ε, που συνιστά προτεραιότητα για την Βελική Προεδρία και εξάλλου σας θυμίζω ότι στο άτυπο Συμβούλιο αναφερθήκαμε σε αυτήν την πρόταση οδηγίας. Κατόπιν θα ήθελα να σας θυμίσω ότι υπάρχει ολόκληρο θεματολόγιο για την αξιοπρεπή εργασία σε συνεργασία με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Ε, διοργανώνουμε και μια κοινή διάσκεψη για αυτό το θέμα της αξιοπρεπούς εργασίας. Ε, αποσκοπούμε σε μια σφαιρικότερη ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα αυτό, χωρίς να ξεχνούμε και το θέμα της ασφάλειας, ε, ψυχοσωματικές διαταραχές, καρκίνος, Κύριε Νταλή, αναφερθήκατε σε όλα αυτά τα ζητήματα. Προφανώς ε, θέλουμε να ενισχύσουμε την προστασία των εργαζομένων, ε, να ενισχύσουμε την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας ε, και προβλέπεται η σχετική συζήτηση στο Συμβούλιο τον Νοέμβριο. Κατόπιν, ε, ε, ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο, μου είπατε, δεν αναφέρθηκα καθόλου στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Απασχόλησης. Μα συνεχώς ασχολούμαι με αυτό, γι' αυτό ίσως και δεν έκρινα χρήσιμο να το αναφέρω. Πρέπει να προσαρμόσουμε αυτό το εργαλείο στα πλαίσια της στρατηγικής 2020. Δεν είναι το μόνο εργαλείο αυτή τη στρατηγική. Το Σεπτέμβρη-Οκτώβρη στην δημοσιονομική αναθεώρηση, στο budget review για το Ευρωπαϊκό αυτό Ταμείο θα δραστηριοποιηθούμε όλος ιδιαίτερως ούτως ώστε να υλοποιήσουμε ε, φιλόδοξες ε, πολιτικές, ε, να προσαρμόσουμε τα κονδύλια και να εξειδικεύσουμε αν θέλετε τη δράση του Ευρωπαϊκού Ταμείου. Κύριε Γιούν, μας μιλήσατε για την οικονομική διακυβέρνηση, μεγάλος αγώνας. Μέχρι στιγμής μας έχουν υποστηρίξει ε, τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο και άρα προχωρούν τα πράγματα. Ε, το θέμα δεν είναι να πείσουμε μόνο το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ε, στο το Συμβούλιο του Οκτώβρη για τη διακυβέρνηση πρέπει να λάβουν σχετικές αποφάσεις. Άρα πρέπει να δραστηριοποιηθείτε και σε επίπεδο κρατών μελών Γεια το Συμβούλιο ΕΕΠΣΚΟ, το Συμβούλιο ΕΜΚΟ θα πρέπει να κάνουν τη μακροοικονομική ανάλυση, να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας βαθμολόγησης, ε, το scoreboard, οι νέοι δείκτες. Χρειάζεται οπωσδήποτε συντονισμός ανάμεσα στις ε, διάφορες επιτροπές και ξέρετε δεν είναι ένας πόλεμος εξουσίας εδώ. Ε, οι, οι δράσεις των μέγεντων δεν είναι συμπληρωματικές. Χρειαζόμαστε μια συντονισμένη προσέγγιση ούτως ώστε σε επίπεδο αγοράς εργασίας να έχουμε την ε, πλέον αποτελεσματική δράση. Ε, πρέπει να υπομιστούμε τις ευθύνες μας ε, ως προς την δημοσιονομική εξυγίανση. Πρέπει να επιστρέψουμε στο 3% αλλά εάν δεν κατοχυρώσουμε τις μελλοντικέ επενδύσεις θα, πέσουμε, θα επαναλάβουμε μάλλον τα λάθη του παρελθόντος ε, και για την οδηγία που μας είπατε για τους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς νομίζω ότι θα γίνει δεύτερος γύρος διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους από πλευρά της Ευρωπαϊκή επιτροπή και θα μας παρουσιάσει ε, η Επιτροπή κατόπιν την ανάλυση της θα μας παρουσιάσει τα πρώτα στοιχεία της ανάλυσης της ήδη στις εκδηλώσεις ε, που οργανώνουμε, διοργανώνουμε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο το, του Δουβλίνου για τη, τους όρους εργασίας. Τώρα, για τις πολιτικές λιτότητες, για το ελάχιστο εισόδημα, το, τον, τον ελάχιστο μισθό, αναφερθήκατε στον ελάχιστο μισθό. Δεν είναι ελάχιστο μισθό, είναι ελάχιστο εισόδημα. Η συνάδελφό μου, η κυρία Αγγελίξ, θα σχολιάσει αυτό το ζήτημα ευθύ αμέσω. Κοιτάξτε, ε, σε επίπεδο ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο Βελγίου το σημαντικό είναι να τονώσουμε την αντιπροσωπευτικότητα των κοινωνικών εταίρων στην όλη συζήτηση που γίνεται για την ε, προσαρμογή της οικονομικής διακυβέρνησης και την υλοποίηση της στρατηγικής 2020. Δηλαδή πώς ε, ακριβώς, ποιος θα είναι ο ρόλος, των, ε, ο νέος προσαρμοσμένος ρόλος των κοινωνικών εταίρων στα πλαίσια της πολιτικής 2020. Σε συνεργασία μαζί τους θα το προσδιορίσουμε αυτό ενώ χαράσουμε τη νέα πολιτική οικονομική διακυβέρνηση. Κυρία Μπιζό, το τέλος δεν νομίζω ότι αυτό είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Χρειαζόμαστε μια σωστή κοινωνική προστασία ε, για όσοι επιζητούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, αλλά θα πρέπει να κινηθούμε και σε επίπεδο ελάχιστου εισοδήματος ε, πρέπει να συνοδεύσουμε τους ανέργους, να τους βοηθήσουμε να ε, επανέλθουν στην αγορά εργασίας. Για την απόφαση στην οποία αναφερθήκατε δεν είναι θέμα ε, δικής μου αρμοδιότητας για την Μπούρκα. για την καταπολέμηση της διακριτικής ε, μεταχείρισης νομίζω είναι θέμα επικουρικότητας, είναι θέμα κρατών μελών. Φυσικά είναι σημαντικό. Ε, κάποια στιγμή θα μπορούσε να ενταχθεί στα πλαίσια της συζήτησης ε, για την οδηγία ε, κατά της διακριτικής μεταχείρισης, αλλά ίσως αρκεί, ίσως να έχουμε ήδη ε, πολλά ζητήματα στο πρόγραμμα της Ευελικής Προεδρίας, αλλά αν το επιθυμείτε μπορούμε να εντάξουμε και αυτό το σημείο στο πρόγραμμά μας. Πρόεδρος, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω εξ ονόματος των συναδέλφων τα καταφέρατε να απαντήσετε τόσο πολλές ερωτήσεις τόσο γρήγορα. Είμαστε αισιόδοξοι ε, για τα επιτεύγματα, τα μελλοντικά επιτεύγματα της Βελγικής ε, Προεδρίας, ε, το προσεχές εξάμεινο. Ε, δυστυχώς δεν ακούσατε όλους τους συναδέλφους, δεν είχαμε χρόνο, αλλά πάντως σας εύχομαι καλή επιτυχία και θα υποδεχτούμε τώρα τρεις από τους συναδέλφους σας. Αντίο.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 Chers collègues, est-ce que je peux vous demander de prendre place euh, à nouveau Παρακαλώ καθίστε και πάλι. De notre matinée s'annonce comme un défi plus grand que la première partie. Το δεύτερο τμήμα συνιστά ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση σε σχέση με το πρώτο. Έχουμε τρεις υπουργούς και μία ώρα στη διάθεσή μας. Συνάδελφοι, υπάλληλοι, θα αναβάλουμε για τις 11 η ώρα την ψηφοφορία για να έχουμε στη διάθεσή μας μία ώρα. Καλωσορίσατε στην σημερινή μας συνεδρία στην αρχή της ε, Βελγικής Προεδρίας. Είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία σας ε, για μας. Έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πρώτη ανταλλαγή. Κύριε Ενκελίνξ, ε, είστε Υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων και Δημόσιας Υγείας. Ο κύριος Μισελ Νταγνά είστε ε, Υπουργό για τις Μεγάλες Πόλεις ε, και κύριε κυρία Ζερζέ είστε Υπουργό αρμόδιος ε, για τα άτομα με αναπηρίες μέσα στο Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων. Je vous Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μα. Ε, κυρία Άγκελεγγ θα πάρει πρώτη το λόγο και κατόπιν οι συναδελφοί σα. Και πριν καν ξεκινήσετε την παρέμβασή σα, έχουν ήδη εγγραφεί οι ομιλητέ στον κατάλογο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Θα... Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριοι Ευρωβουλευτέ το πακέτο μέτρων για την απασχόληση της καταπολέμησης της κρίσης της ανεργίας διεξοδικά το, το έχετε εξετάσει. Υπάρχει όμως και ένα επιπλέον σημείο στο οποίο θα έπρεπε να συνεργαστούμε. Συνολικά δηλαδή το θέμα της κοινωνικής συνοχής. Είχαμε ένα άτυπο συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα, Συμβούλιο Υπουργών, και οι Υπουργοί τι διαπίστωσαν. Διαπίστωσαν ότι η οικονομική και η κοινωνική κρίση, η χρηματοοικονομική κρίση έχει τρομερές επιπτώσεις επειδή η ανεργία αυξάνεται εκρηκτικά, η επισφαλής εργασία και η επισφαλής κατάσταση των εργαζομένων αυξάνεται και εδώ διακυβεύεται όχι μόνο ο παραδοσιακός ρόλος της ευημερία, αλλά πρέπει να δημιουργηθεί μια σπίδα ώστε να μπορέσουμε να προστατέψουμε τους πολίτες μας από αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις. Διαπιστώσαμε ότι ήταν επικίνδυνο σε σχέση με τους, ε, τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών τώρα στην Ευρώπη να καταλήξουμε σε ένα κοινωνικό ανταγωνισμό, διότι αυτό θα υποβάθμιζε και θα αποσταθεροποιούσε τις ισορροπίες των κοινωνικών εταίρων και θα υπονόμευε τις ε, σχέσεις. Ε, είπαμε ότι είναι σημαντική η μακροοικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και έχω τη βεβαιότητα ότι η συνάδελφος σας εξέθεσε τα σχετικά διεξοδικά από κοινού μαζί σας θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα μέσα, τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για την επίτευξη τη στρατηγική του 2020. Έχουμε αριθμητικά μεγέθη παράλληλα με την απασχόληση. Έχουμε αυτές τις, αυτά τα μεγέθη και θέλουμε να προσπαθήσουμε με τη βοήθεια αυτών των μέσων να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια. Έχουμε και την οδηγία, την οδηγία ε, 10, την οδηγία C έχουν βελτιωθεί τα πράγματα όσον αφορά τις ε, εργασίες και από πλευράς της Κοινοβουλευτικής σας Επιτροπής. Από τον προηγούμενο Ιούνιο έχουμε βελτιώσει το κείμενο με βάση τις συζητήσεις ε, που έγιναν από πλευρά σας και φαίνεται ότι μπορεί να δοθεί συνέχεια με βάση αυτή την καλή συνεργασία να προαχθούν αυτά τα θέματα μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Συμβουλίου ιδιαίτερα σε τρία σημεία σε τρία θέματα που είναι πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Δεν έχει ολοκληρωθεί η εργασία, αλλά έχει τονιστεί μέσα στο πλαίσιο αυτό ότι θα πρέπει να λάβουμε ιδιαίτερα την αηφορία στην χρηματοδότηση όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά από πλευράς των κρατών μελών θα πρέπει να προαχθεί αυτή η παράμετρος ώστε να προαρθούν οι θετικές πτυχές και επιπτώσεις ε, μέσα στο πλαίσιο και των εθνικών προϋπολογισμών σε σχέση με τους ε, εργαζόμενους και όταν μειώνεται η φτώχεια είναι σημαντικό να έχουν μεγαλύτερο εισόδημα οι πολίτες και να ανακουφιστούν όσον αφορά τις φορολογικές επιβαρύνσεις και να υπάρχει η δυνατότητα μέσω δημόσιων επενδύσεων και υπηρεσιών να τονωθεί η κατάσταση. Είναι ένα παράδειγμα που μπορεί να βρεθεί ένα άνοιγμα, μια αφετηρία ώστε να ξεκινήσουμε οι προτεραιότητες αυτές να αρχίσουν να εντάσσονται μέσα σε αυτή την οδηγία 10. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ο οδικό χάρτης ε, για την πορεία που θα ακολουθήσουμε. Roadmap, ε, ο οδικός χάρτης για μας, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το κοινωνικό χάσμα και να προχωρήσουμε στη στρατηγική 2020. Και στο άτυπο συμβούλιο έχουμε επίσης και μία εντολή αυτή την κοινωνική προστασία ή την Επιτροπή για την Κοινωνική Προστασία να ζητήσουμε να υποβληθούν ε, δείκτες για την υλοποίηση της οδηγίας 10. Και επίσης ζητήθηκε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υπάρξει η αντίστοιχη ναυαρχίδα ως εγχείρημα, ως πρωτοβουλία για να καταπολεμηθεί η φτώχεια. Αυτή η ναυαρχίδα, αυτό το πρόγραμμα ε, δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της Οδηγίας 10 την οποία θα υποστηρίζει και θα προάγει. Πρόκειται για το θέμα ακριβώς της κοινωνικής συνοχής ε, συνολικότερα. Κατά την Προεδρία του Συμβουλίου, εμείς τονίσαμε ως Βελγική Προεδρία ότι η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού έχει μεγάλη σημασία για μας. Μια διάσκεψη θα ασχοληθεί τον Σεπτέμβριο του 2010 ακριβώς με αυτό το θέμα και θέλαμε στη συνέχεια να τονίσουμε εξάλλου πόσο σημαντικό είναι το άρθρο 9 της Συνθήκης Λισαβόνας, η περιβόητη αυτή κοινωνική ρήτρα. Και θα πρέπει να γίνει γνωστότερο αυτό. Και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από καιρούς καιρών για αυτό τον τομέα εκπονείται κάποια πρόταση. Θα πρέπει όμως να υπάρχει διαφάνεια σε σχέση με αυτό το θέμα ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα σε σχέση με την οδηγία επαριθμό 10. Όπως είπα για τις υπηρεσίες ε, ο, καθολικού συμφέροντος ε, θα πρέπει να λάβουμε αυτό το σημείο ιδιαίτερα υπόψη. Στην Ευρώπη διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο και το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο δεν προσαρμόζεται σωστά, δεν είναι το πιο ενδεδειγμένο και κατάλληλο για να προβούμε στην τόνωση αυτών των υπηρεσιών. Συζητήσαμε με τους stakeholders, με τους εμπλεκόμενους ε, και κατά τη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας δύο θέματα θα εξεταστούν. Πρώτον θα προσπαθήσουμε να ε, καταρτήσουμε ένα πρόγραμμα δυνατοτήτων για να προσαρμοστούμε σε αυτές τις δράσεις και θα βασιστούμε στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και επίσης θα ε, δραχθούμε της ευκαιρίας ε, ώστε οι εργασίες της Επιτροπής για την Κοινωνική Προστασία να χρησιμοποιηθούν ώστε να υπάρξει η τόνωση αυτού του πλαισίου. Αυτά σε σχέση με το πλαίσιο αυτό και την ποιότητα που θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με αυτόν τον τρόπο και θα έχουμε και ένα τρίτο φόρουμ το οποίο και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον τον Οκτώβριο αυτό το φόρουμ. Το φόρουμ αυτό θα ασχοληθεί και με το να προπαρασκευάσει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που θα ακολουθήσει μετά Αυτά είχα να πω. Θα δώσω τον λόγο συναδέλφου. Euh, euh, euh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Από πλευρά μου, εξ μου και εξ των συναδέλφων μου, θα ήθελα να πω σύντομα δύο λόγια για την φτώχεια και για τα άτομα με ε, ειδικέ ανάγκες. Κατά τη διάρκεια αυτής της ε, δική μα προεδρία. Ολοκληρώνεται και λίγη το έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας. Πολύ σημαντικό ορόσημο αυτό. Στην Λισαβόνα είχαμε φιλόδοξους στόχους που διατυπώθηκαν ώστε να καταπολεμηθεί η φτώχεια, να ξεριζωθεί η φτώχεια. Δυστυχώς όμως δεν καταφέραμε να πετύχουμε αυτό το στόχο. Και σίγουρα θα απαιτηθεί να υπάρξουν περαιτέρω εργασίε και μεθοδολογικά. Όσον αφορά το Βέλγιο και την Προεδρία μα, θα ήθελα να αναφέρω τα εξή σημεία. Πρώτον, το ελάχιστο εισόδημα. Και αυτό είναι φυσικά ένα σημαντικό σημείο, διότι το πιο σημαντικό είναι φυσικά η τα κατάλληλα εισοδήματα που θα διασφαλίζονται για τα άτομα που βρίσκονται ε, και προς, ε, κοντά στο περιθώριο. Δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα με ένα 75% ε, του μέσου εισοδήματος να τονωθεί αυτή η πτυχή. Το δεύτερο θέμα είναι η καταπολέμηση της φτώχειας των παιδιών. Είναι ένα σφαιρικό θέμα αυτό ε, όπου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη θέματα της πρόσβασης παιδιών και οικογενειών ε, σε ε, υπηρεσίες. 20% ζουν κάτω από την, το επίπεδο της φτώχειας. Θέλουμε να ξεκινήσει μια ευρωπαϊκή συζήτηση για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. Και εδώ φυσικά πρόκειται επίσης και για στόχους μείωσης ακριβώς, για ένα στόχο μείωσης της φτώχειας που ε, πλήττει τα παιδιά. Αυτό αφορά και τα δικαιώματα των παιδιών, αλλά είναι ένα πρόβλημα που έχει πολλές επιτυχές και είναι σύνθετο και αφορά και τα θέματα στέγασης και την συμμετοχή στην κοινωνική ζωή και θέματα υγείας. Όλες αυτές οι παράμετροι διαδραματίζουν ένα ξεχωριστό ρόλο μέσα σε αυτό το σύνολο. Ένα τρίτο θέμα είναι το ζήτημα των αστέγων και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί μια συνενετική συνδιάσκεψη θα διεξαχθεί υπό την Βελγική Προεδρία και μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στις 18 και 19 Δεκεμβρίου θα λάβει χώρα ώστε οι συστάσεις ε, να, για την ε, ένταξη αυτών των ατόμων να εκπονηθούν. Δηλαδή να δημιουργηθεί μια, ε, ένας χώρος εργασίας, μια αγορά εργασίας που θα παρέχει δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες για αυτά τα άτομα. Και με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών θα διεξαχθεί αυτό το φόρουμ και θα επισημανθεί και θα αναφέρεται πόσο σημαντικό είναι να επενδύσουμε στην κοινωνική οικονομία της αγοράς και στις κοινωνικές υπηρεσίες Όσον αφορά τα άτομα αυτά, τα άτομα με ειδικέ ανάγκε, θα πρέπει ο μύτο τη Αριάδνη να είναι η υλοποίηση του, των αρχών των Ηνωμένων Εθνών και του προγράμματο αυτού για τα άτομα με ειδικέ ανάγκε. Είναι μια σημαντική πρόοδο, παγκόσμια αυτή, ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε αυτέ τι αρχέ, εχει Έχει προσυπογραφεί από αρκετά κράτη-μέλη μέχρι σήμερα και με τι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε από κοινού να μεριμνήσουμε για την υλοποίηση ενεργοποίηση αυτών των αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό να γίνει φυσικά σε συνεργασία με κάθε ένα κράτος μέλος ξεχωριστά διότι στο τέλος τέλος πρόκειται εδώ για το δικαίωμα των ανθρώπων, των ατόμων αυτών να είναι πολίτες και μάλιστα πλήρεις πολίτες της κοινωνίας μας και να έχουν δυνατότητες πληροφόρησης, προσπελασιμότητα στις υπηρεσίες, πρόσβαση στα κτίρια, όπως και δικαιώματα που έχουν οι άλλοι πολίτες εξάλλου και είναι αυτονόητα για αυτούς. Και γι' αυτό στις 18 και 19 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί μια συνδιάσκεψη, όπως είπα, ώστε να συζητήσουμε για την εφαρμογή, την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας των Ηνωμένων Εθνών, Εθνών υπό τη συμμετοχή φυσικά των ατόμων με ειδικέ ανάγκες. Και ελπίζουμε ακριβώς να υπάρξει μεγάλη συμμετοχή των ατόμων με ειδικέ ανάγκες θα υπάρξει μια ανταλλαγή απόψεων για τι βέλτιστε πρακτικέ για να δούμε πώ τα κράτη-μέλη αυτά τα δικαιώματα υλοποιούνται και είναι σεβαστά σε ανοιχτή συζήτηση με του ενδιαφερόμενου και κατά την δεύτερη ημέρα θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των κρατών μελών και των κρατικών αρχών των κρατών μελών. Και θα πρόκειται για όλα τα επίπεδα, από το τοπικό μέχρι το περιφερειακό, το εθνικό και το ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα σημαντικό θέμα είναι και ο δεοντολογικό κώδικα, Με άλλα λόγια δηλαδή, θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει το επιμερισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και του ευρωπαϊκού επίπεδου από την άλλη πλευρά. Και θα καταβάλουμε προσπάθειες με αυτό το, μέσα σε αυτό το πλαίσιο αυτούς τους προβληματισμούς ενεργά να τους ε, προωθήσουμε όσον αφορά την ε, ε, θέσπιση ενός διοντολογικού κώδικα και την δημιουργία ενός πρωτοκόλου που θέλουμε με τα κράτη-μέλη και αυτό να προωθεί ώστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να τύχει συνέχεια σε αυτό το εγχείρημα. Χαιρετίζουμε επίσης τις εργασίες της Ισπανικής Προεδρίας. Σε 7 Ιουνίου 2009 στο Λουξεμβούργο υιοθετήθηκε το νέο πλαίσιο για τις αναπηρίες, όπου αναφέρεται με ποιο τρόπο σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να έχουμε μια πολιτική όπου θα εντάσσονται τα άτομα με αναπηρίες, θα εφαρμοστεί ένα mainstreaming για αυτά τα άτομα με αναπηρίες, ώστε να μπορέσουν ε, να συμμετάσχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο κρατών μελών ε, για την προστασία των ατόμων που πάσχουν από αναπηρίες. Ε, τέλος, οδηγία για την κατάργηση της διακριτικής μεταχείρισης. Ε, φυσικά αυτό υπερβαίνει το πεδίο αρμοδιοτήτων της κυρίας Μελκέ που ήταν πριν από μας στο βήμα της Επιτροπής σας. Ε, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί, γίνεται έντονος διάλογος, περιμένουμε όμως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλιώς δεν μπορούμε να προοδεύσουμε ε, για κάποια σημεία, κυρίως για όσους πλήττονται από τις αναπηρίες, αυτό που μας απασχολεί δηλαδή, αλλά όχι μόνο, ε, όλος ιδιαίτερος για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στον τομέα ε, της καταπολέμησης διακριτικής μεταχείρισης ε, κατά των ατόμων με αναπηρίες. Ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Νταχτάν θα πάρει το λόγο ε, για πέντε λεπτά. Ίσως μπορείτε να μας πείτε αν στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου κάποια στιγμή έχει προβλεφθεί το θέμα της πράσινης βίβλου που μόλις επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πότε θα συζητηθεί αυτό το θέμα. Ε, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους Γάλλους ε, συναδέλφους ε, γιατί σήμερα είναι εθνική εορτή. Στις 7, 8 και 9 Ιουλίου στο άτυπο συμβουλίο συζητήθηκαν πολλά από αυτά τα ζητήματα και από ό,τι κατάλαβα ε, στο θέμα των μεταρρυθμίσεων ε, η λέξη κλειδί είναι η επικουρικότητα. Από ό,τι κατάλαβα, η, η πράσινη βίβλος ε, βασίζεται στις ε, κοινέ εργασίες της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας ε, και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Υπάρχουν 14 βασικά ζητήματα σε αυτό το διάλογο. Ε, στον λογοέγγραφο τονίζονται μεταξύ άλλων η ανάγκη της οικονομικής ανάκαμψης, ε, της δημοσιονομικής εξυγίανσης, ε, ανάγκη κατοχύρωσης παρκούς επίπεδου για τις συντάξεις, αύξηση των, του συντάξιμου ορίου, ηλικιακού ορίου ρύθμιση των κεφαλαιοποιητικών ε, συνταξιοδοτικών συστημάτων, ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών, αυξανόμενος ρόλος ε, των συνταξιδοτικών ταμείων, θεωρώ ότι κάθε κράτος μέλος βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του θα πρέπει να ρυθμίσει όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά υπάρχει και το θέμα ε, της μεταφοράς ε, των συντάξιμων δικαιώματων για τις επικουρικές συντάξεις των διασυνοριακών εργαζομένων, ε, της φερεγγιότητας των συνταξιοδοτικών ταμείων, της κοινοποίηση των πληροφοριών ή των στατιστικών στοιχείων. Νομίζω ότι αυτά μπορούν να αποτελέσουν ένα αντικείμενο ενός κανονισμού ή μιας οδηγίας. Ε, οφείλουμε να προβληματιστούμε για αυτά τα 14 σημεία της Επράσινης Βίβλου, κυρίως όμως ε, για την βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Γνωρίζω ότι αυτό θα είναι το βασικό σημείο της υπουργική διάσκεψης που θα γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου στη Λιέγη για το μέλλον των συνταξιδοτικών συστημάτων η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας και η Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής φυσικά θα συνεργαστούν με τη Βελική Προεδρία. Ε, σε αυτό θα συμμετάσχουν και οι πολίτες, ούτω ώστε ευελπιστούμε να συνταχθεί η Λευκή Βίβλος για τις συντάξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και από αυτή την άποψη είναι απαραίτητο κατά τη γνώμη μου να προβληματιστούν ε, ταυτόχρονα και τα Συμβούλια Εκοφήν και ΕΠΣΚΟ για αυτό το θέμα και οι συντάξεις είναι ένα μόνο σημείο, βέβαια πάρα πολύ σημαντικό, για την καταπολέμηση της στόχης στην οποία προαναφερθήκατε, ε, αλλά επίσης επιτρέπει στους πλέον ε, ηλικιωμένους, στους ε, πρεσβυτέρους της κοινωνίας μας να, να έχουν πρόσβαση σε μια αξιοπρεπή γύρανση. Ευχαριστούμε κύριε Βερντά. κυρία Ιάκαν Σαρή και ο κύριος Γιούρη θα πάρουν πρώτοι το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα πράγμα δεν είναι απόλυτα σαφές πλέον για μένα και πρέπει να το αναφέρω αυτό. Και αυτό είναι πώς η Βελγική Προεδρία σκέφτεται, τι έχει υπόψη τη και τι θα κάνει σε σχέση με την οδηγία περί εργαζομένων. Πώς θα την αντιμετωπίσει. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για την Ένωση η ελευθερία κυκλοφορίας και είναι ένα σημαντικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι δεν είναι. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν τα σχετικά. Η ελευθερία κυκλοφορίας όμως έχει οδηγήσει και σε εχθρότητα προς τους ξένους, σε ξενοφοβία και εχθρότητα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να ξέρω τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την οδηγία περί εργαζομένων. Και δεύτερον, δεύτερον ακριβώς τίθεται εδώ το θέμα των ελάχιστων μισθών ή του ελαχίστου εισοδήματος. Ελπίζω, πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές ασάφειες εδώ. Θα πρέπει πρώτα οι ορισμοί να καθοριστούν. Να καθορίσουμε και να πούμε τι είναι εκείνο το οποίο η Βελγική Προεδρία θέλει να πετύχει όσον αφορά αυτό το θέμα. Ελάχιστο μισθό θέλει να πετύχει ελάχιστο εισόδημα. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ ο κύριος και ο κύριος Κομφεράτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους, ε, την Υπουργό και τους Υφυπουργούς ε, για τις ε, παρουσιάσεις του. Δεν έχω πολύ χρόνο, οπότε θα ήθελα ευθύς αμέσως να αναφερθώ στις ε, προτεραιότητες ε, της Βελγικής και Ουγγρικής Προεδρίας. Ε, μία από αυτές τις προτεραιότητες είναι η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. Αυτό που θα πρέπει να διαπιστώσουμε είναι αν δυνάμεθα να ποσοτικοποιήσουμε το πρόβλημα για να έχουμε απτά αποτελέσματα και μια παρακολούθηση του ζητήματος μελλοντικά. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Κομφεράτη και η κυρία Λίν. Σα ευχαριστώ. Πολύ συχνά στην εργασία μας εδώ γίνεται λόγος για αξιοπρεπή εργασία των είναι η αξιοπρεπής εργασία, εκείνη η μορφή εργασίας όπου τα δικαιώματα των εργαζομένων αναγνωρίζονται, είναι σεβαστά και στις χώρες τους ε, επιπλέον, επιπλέον πέρα από το κοινοτικό ε, δίκαιο ε, προβλέπονται και συλλογικές συμβάσεις και σωστή αμοιβή της εργασίας. Τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Είναι αρκετά διαδεδομένο να υπάρχουν και κάποια αρνητικά φαινόμενα. Με άλλα λόγια, άτυπη εργασία ή επισφαλής εργασία. Εκείνοι οι πολίτες δηλαδή που είναι πολίτες των χωρών αυτών και που ασκούν μια δραστηριότητα που όμως η αξιοπρέπειά τους ε, και δεν αναγνωρίζεται και η εργασία δεν είναι αξιοπρεπής. Δεν ισχύουν συλλογικέ συμβάσεις, δεν ισχύουν σωστές ε, δίκαιες αμοιβέ και ένα άλλο φαινόμενο είναι η παράνομη εργασία. Είναι η περίπτωση ανθρώπων που έχουν γεννηθεί αλλού, έρχονται εδώ να εργαστούν, αλλά και για αυτούς ε, δεν υπάρχει κανένα είδος προστασία που να διασφαλίζεται στην εργασία που επιτελούν, ούτε μέσω συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέσω εργασιακών διατάξεων και πρέπει να, αποτελε... να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά αυτά τα φαινόμενα. Θέλω να ξέρω, θα γίνει κάτι από την ε, Βελγική Προεδρία. Δεν πρόκειται μόνο για την αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων, αλλά και για τις προοπτικές τους. Δεν έχουν ε, καθόλου δικαιώματα να εισπράξουν, να τους καταβληθεί μια σύνταξη ή να απολαύσουν δικαιώματα από την εργασία τους. Είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η κατάσταση και είναι κάτι το οποίο έχει οξυνθεί τώρα κατά τη διάρκεια της κρίσης και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Euh, Ευχαριστούμε. Η κυρία Λίνε και ο κύριος Μπακ. Ευχαριστώ. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία αναφέρατε. Θα αναφερθώ σε κάποια από αυτά. Κύριε Όγκελινγκ, αναφέρατε σε σχέση με τι ε, φτωχότερες χώρες και για την βελτίωση αυτών των πραγμάτων. Προφανώ όλοι γνωρίζουμε ότι δεν ε, λειτουργήσαν ε, σωστά κάποια πράγματα στο παρελθόν. Όμω πώ βλέπετε ότι μπορούν να βελτιωθούν κάποιε πτυχέ ιδιαίτερα όσον αφορά την καταπληκτική καταπολέμηση της φτώχειας, την αντιμετώπιση των θεμάτων των αστέγων. Έχετε κάτι υπόψη μακροπρόθεσμα σε σχέση με... Ε, εγώ ασχολούμαι με ένα διοντολογικό κώδικα, θα ήμουν ευγνώμων αν μου δίνατε κάποιες απόψεις από πλευρά, από πλευρά σας. Όσον αφορά το ελάχιστο εισόδημα, πάλι έχουμε το πρόβλημα. Κάποιος ανέφερε ότι χρησιμοποιείται ο όρος ελάχιστος μισθός, άλλοι αναφέρουν το ελάχιστο εισόδημα. Εγώ επικεντρώνομαι στο ελάχιστο εισόδημα. Δηλαδή όχι ε, καθαρά καθαρά μέσω της απασχόλησης αλλά και μέσω της κοινωνικής ασφάλισης κυρίως. Θα ήθελα τις απόψεις σας επί αυτού του θέματος για το ελάχιστο εισόδημα. Αν θα έπρεπε ένα ελάχιστο εισόδημα να ισχύει για όλες τις χώρες μέλη, πράγμα το οποίο εγώ πιστεύω ε, ότι θα έπρεπε να γίνει, αλλά μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και ίσως ε, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του ανοιχτού συντονισμού και πάλι για την οδηγία για τα άτομα με ειδικές ε, ανάγκες η τροχοπεδίθηκε στο Συμβούλιο αυτό το θέμα και χάρηκα που άκουσα ότι αναφέρατε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για άτομα με ειδικέ ανάγκε. Έχετε κάποια προγράμματα ή σχέδια για να προσπαθήσετε να ασκήσετε πίεση σε εκείνα τα κράτη-μέλη που δεν έχουν προσυπογράψει ή κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, διότι φυσικά έχει τεράστια σημασία. Κάθε ξεχωριστό κράτο μέλο αυτή τη φορά να μπορέσει να επικυρώσει και να ε, εγκρίνει αυτή τη σύμβαση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπάκη, η κυρία Καστέξ. Äh, Θα ήθελα ε, να μας μιλήσετε λιγάκι για τον συντονισμό των διαφόρων πολιτικών. Ο κύριος Νταρντέν πολύ σωστά επισήμανε ότι η οικονομική ανάπτυξη, η ε, κοινωνική πολιτική, η αγορά εργασίας είναι ε, τρία διαφορετικά θέματα και παρότι η συζήτηση για το με την πράσινη βίβλο περί συντάξεων βρίσκεται τη γενέστη, αλλά παρόλα αυτά ο στόχος είναι να ε, υπάρχει περισσότερος χρόνος εργασίας. Και διερωτώ με πώς αυτό μπορεί να συμβιβαστεί με την εργασία μέχρι τις ηλικίε περίπου των 70 ετών. Αυτή τη στιγμή έτσι και αλλιώς ε, στην αγορά εργασίας οι άνω των 50 ετών έχουν πρόβλημα να βρουν νέα θέση απασχόλησης. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι η πολιτική αυτή δεν είναι συνεπής. Κατά τα άλλα, θα ήθελα σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη, εγώ να σας επισημάνω τα μέτρα λιτότητας, τα οποία έτσι και αλλιώ θα πλήξουν τους κοινωνικά ασθενέστερους. Και τελικά, αντί να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και να την περιορίσουμε, εγώ θεωρώ ότι θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, θα έχουμε περισσότερους πέννητες. Κατά τα άλλα, θα ήθελα να σας ε, επισημάνω το θέμα των ατόμων με αναπηρία, τα δικαιώματα των επιβατών ε, στα λεωφορεία. Σε αυτό το θέμα δεν συμφωνήσαμε. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να σας παρακαλέσω μέσω της διαιτησίας να επιμείνετε έτσι ώστε πράγματι να βρούμε μια λύση. Ευχαριστώ, Madame Castex, puis Ευχαριστώ η κυρία Καστέξ. Ε, Υπουργέ, μία ερώτηση για τις υπηρεσίες κοινή ωφελίας διοργανώσετε το τρίτο φόρουμ για τις κοινωνικές ε, υπηρεσίες, αλλά πέραν αυτού έχετε μία ε, πρωτοβουλία ε, νομοθετικού χαρακτήρα, δηλαδή να εκπονήσετε μία χάρτα ποιότητας, επιθυμείτε να δημιουργήσετε, θα σας υποστηρίξουμε εμείς, επιθυμούμε. αυτή η όθηση που θα δώσετε, που ελπίζουμε να δώσετε σε αυτό το θέμα, να έχει και κάποια συνέχεια ευελπιστούμε ότι ε, το Συμβούλιο σταθερά θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα, ούτω ώστε να κατοχυρώσει τις υπηρεσίες ε, κοινή ε, ωφελίας. Γνωρίζετε ότι στην Επιτροπή μας συζητούμε αυτό το θέμα. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ε, εξασφαλίσουμε ε, την καθολική πρόσβαση ε, και να κατοχυρώσουμε τον καθολικό χαρακτήρα αυτών των υπηρεσιών αποφεύγοντας έτσι αυτές οι υπηρεσίες να αφορούν μόνο τις εξαιρετικά μενεκτούσες πληθυσμιακές ομάδες. Ευχαριστούμε η κυρία Ντελή. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Καλημέρα και σας ευχαριστούμε που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Θα ολοκληρώσετε το έτος κατά πολέμηση φτώχειας ε, και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ξέρετε, ε, ε, έχω ξαναθέσει αυτό το ερώτημα, αλλά στη συνάδελφό σας. Λοιπόν, προτίθεται η Βελική Προεδρία να υποστηρίξει μια πρωτοβουλία για να θεσπιστεί η περίφημη οδηγία πλαίσιο για το ελάχιστο εισόδημα. Κατόπιν, φορολογία υψηλών εισοδημάτων. Αυτό θα μπορούσε να μας βοηθήσει στην δημοσιονομική εξυγίαση και την εξυγίαση της κοινωνικής ασφάλισης. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να ε, ξεκινήσουμε τι εργασίε προ αυτή την κατεύθυνση και να ε, έχουμε προληπτική δράση για τη φτώχεια. Είναι βασικό στοιχείο. Για του αστέγου. η στέγαση δεν είναι συνιστά αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ είναι εφαρμοστεί η αρχή τη Επικουρικότητα. Με ποιο τρόπο λοιπόν εσείς θα ασκήσετε πίεση στα κράτη-μέλη, ούτω ώστε να σεβαστούν το ότι κάθε Ευρωπαίος πολιτή δικαιούται πρόσβαση σε μια αξιοπρεπή στέγη ε, και με το, για τους αστέγους. Υπάρχουν πολλοί άριθμες δηλώσεις ε, Πρόσφατα η κυρία Λίν, η κυρία Φιγκυρέιτο και άλλοι συνάδελφοι ε, προσπέγραψαν μια σχετική δήλωση. Ωραία, εγώ θέλω να ξέρω ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσετε για να ασκήσετε πίεση. Δεν μπορείτε να περιμένετε το 2015. Υπάρχουν άστεγοι που πεθαίνουν κάθε χρόνο. Ευρωπαίοι πολίτε πεθαίνουν κάθε χρόνο. Δεν μπορούν να περιμένουν να λήξει το έτος της καταπολέμησης τη φτώχεια. Ε, ευχαριστούμε. Νομίζω θα ευνοηθεί η σοσιαλιστική ομάδα, ε, αλλά όλοι μου έχουν ζητήσει το λόγο. Δεν φταίω εγώ. Θα προσπαθήσουμε να τους ακούσουμε όλους τους συναδέλφους. Ο κύριος Ντερόζα. Ε, uh, σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ κύριε Υπουργή για την παρουσίασή σας σήμερα το πρωί. Την ερώτησή μου προς Όγκελεγκ που συσχετίζεται με το ίδιο θέμα που έθεσε και η κυρία Καστέξ με το κοινωνικό πλαίσιο των υπηρεσιών ε, κοινού συμφέροντος. Είμαι εισηγητής για το μέλλον των υπηρεσιών κοινού συμφέροντος ε, και σε σχέση με την Βελγική Προεδρία παρακολούθησα το σεμινάριο εχθές για τις τεχνικές πτυχές του θέματος. Πρέπει να πω ότι ήταν ένα εξαιρετικό σεμινάριο και σας συγχαίρω για την διοργάνωσή του. Ήταν ε, πραγματικά άξιζε τον κόπο, άξιζε τον τεράστιο κόπο και προσπάθεια που επενδύθηκε γι' αυτό. Ερώτησή μου, όταν λέτε ότι το νομικό πλαίσιο δεν αντιμετωπίζει το θέμα του πώς οι υπηρεσίες γενικού συμφέροντος θα διοργανώνονται. Στόχος σας είναι να χρησιμοποιήσετε το άρθρο 14 των συνθήκων για να επιληθεί, να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα του νομικού πλαισίου ή μήπως ε, εξετάζετε άλλες πτυχές και παραμέτρους όσον αφορά το νομικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα όσον αφορά θέματα ανταγωνισμού και θέματα δημόσιων αγορών ή προμηθειών. Και όσον αφορά το θέμα της επικουρικότητας επίσης το γεγονό ότι οι γενικέ υπηρεσίες, κοινωνικές υπηρεσίες ε, κοινού συμφέροντο δεν υφίστανται στα κράτη-μέλη εκτό αν αποφασίσουν ότι θα παρέχονται τα ίδια τα κράτη-μέλη. Δεν είναι θέμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να το αποφασίζει αυτό. Είναι θέμα περίπλοκης σύνθεση, πώ θα διοργανώνονται και θα πληρώνονται και θα καλύπτονται τα κόστη αυτών των υπηρεσιών. Και έχουμε εδώ και τα θέματα των ε, επιχορηγήσεων, των κρατικών ενισχύσεων ε, και των θεμάτων ανταγωνισμού. Όλα αυτά θα πρέπει σφαιρικά να αντιμετωπίζονται αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί ότι οι υπηρεσίες κοινωνικού συμφέροντος, οι κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος θα θέλουμε να επιβιώσουν και ε, να μην ε, απαλληθούν, γιατί βλέπουμε ότι δίνουν αγώνα επιβίωσης. Ευχαριστώ. Ο κύριο Νταχντά. Ευχαριστώ. Δεν θα καταχραστώ το χρόνο, γιατί ξέρω ότι δεν έχουμε και πολύ στη διάθεσή μας. Κάποια σύντομα σχόλια. Χαίρομαι πάρα πολύ για τις ε, πρωτοβουλίες που ανακοίνωσαν ε, οι διάφοροι υπουργοί για όλα αυτά τα ζητήματα που μας απασχολούν, ούτω ώστε να γίνει πιο ε, κοινωνική η Ευρώπη μας, να έχει ένα εντονότερο κοινωνικό πρόσωπο. Όπως είπε και η κυρία Ένκολίξε και η κυρία Μιλκέ, ε, το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ θα πρέπει να συνεργαστεί για την καθοδήγηση πολιτικής 2020 και για την ε, προώθηση της μεταρρύθμισης της οικονομικής διακυβέρνησης. Θέλω να επανέλθω σε μια πρωτοβουλία που προαναφέρθηκε, η καταπολέμηση της φτώχειας. Αυτή με απασχολεί. Πολλοί συνάδελφοι ε, σχολίασαν αυτή την πρωτοβουλία ήδη. Εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι ε, για να επιτύχουμε τους στόχους, ε, για να σημειώσουμε πρόοδο, πρέπει να ποσοτικοποιούμε τους στόχους, αλλά πρέπει και να τους υλοποιούμε. Τα κράτη λοιπόν θα πρέπει συγκεκριμένα να υλοποιήσουμε τους στόχους. Πώς θα γίνει αυτό. Μας μιλήσατε ήδη για τους δείκτες. Ε, οι δείκτες είναι ένα στοιχείο κλειδί για την υλοποίηση των μέτρων. Και όπως είπε και η κυρία Λίν και η κυρία Ντελή, άλλο ένα σημαντικότατο στοιχείο είναι το ελάχιστο εισόδημα. Είναι σημαντικό κατ' εμέ να οδηγηθούμε σε μια νομοθετική πρωτοβουλία ούτως ώστε να έχουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο που θα ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη, να έχουμε ένα ελάχιστο εισόδημα, είναι ένα ελάχιστο πρότυπο, αν θέλετε, ε, το οποίο πρέπει να επιδιώξουμε. Ευχαριστούμε, η κυρία Πλόμπ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους Υπουργού ε, για τις εισηγήσεις τους και εύχομαι κάθε επιτυχία στη Βελγική Προεδρία. Δύο ερωτήσεις. Η καταπολέμηση της φτώχεια. ακριβώς τη φτώχεια των παιδιών Κύριε Υπουργέ, το, πέρυσι είχε εγκριθεί ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπου πρόκειται για την κατάσταση των παιδιών που παραμένουν μόνα τους στο σπίτι και εργάζονται οι γονείς τους στην Αλοδαπή. Θα ήθελα να σας ερωτήσω αν από πλευρά της Βελγικής Προεδρίας έχετε υπόψη σας να αναλάβετε μια πρωτοβουλία ακριβώς όσον αφορά τις συστάσεις που διατύπωσε τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του πέρυσι. Πρώτη μου ερώτηση αυτή. Δεύτερη ερώτηση προς τον κύριο Νταρντέν. Και εδώ πρόκειται ακριβώς ε, για το σύστημα των συντάξεων, συνταξιοδοτικό σύστημα και την βιωσιμότητά του, την αηφορία του. Κύριε Υπουργέ, ζούμε όλοι σε μια οικονομική, χρηματοοικονομική κρίση και όλο αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στον κοινωνικό τομέα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι πολλοί άνθρωποι μεταξύ 45-50 ε, ετών έχουν χάσει την θέση εργασίας τους και στην αγορά εργασίας υπάρχουν μεγάλα εμπόδια για αυτά τα άτομα να βρουν μια νέα απασχόληση. Υπάρχει μια έννοια, η έννοια της ε, ε πρώιμη συνταξιοδότηση. Θα ήθελα από πλευρά σα, κύριε Υπουργέ, που ασκείτε τώρα την Προεδρία του Συμβουλίου από πλευρά του Βελγίου, να ξέρω αν έχετε μια προσέγγιση για αυτό το θέμα, για την έγκαιρη ε, πρώιμη συνταξιοδότηση. Επειδή ακριβώ στα κράτη-μέλη υπάρχουν τεράστιε διαφορέ. Ε, κάποιοι λένε είναι θετικό, λέει αυτό το μέτρο. Καλό είναι το συνταξιοδοτικό σύστημα να χρησιμοποιήσει μια τέτοια δυνατότητα να καταπολεμηθεί η φτώχεια και να έχουν οι άνθρωποι μια ευκαιρία στη ζωή του. Άλλοι όμω λένε ότι η πρώιμη συνταξιοδότηση είναι κάτι αρνητικό, είναι κάτι μάλλον το οποίο έχει αρνητικές επιπτώσεις για την κοινωνική ασφάλιση. Σας ευχαριστώ θερμά για την απάντηση των ερωτήσεών μου προημίου και εύχομαι κάθε επιτυχία. Θα έλεγα επίσης ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη το συσχετισμό της εντολής σας και το έργο του κυρίου Φαν Ρόμποϊ, που είναι η χέγγια ακριβώς για επιτυχή Βελγική Προεδρία. Ευχαριστώ. Merci. Σας ευχαριστώ. Πριν σας ξαναδώσω το λόγο και στους τρεις, θα ήθελα και εγώ να ανασχολιάσω την αναφορά που κάνατε στο άρθρο 9. Προφανώς όταν μιλάμε για την εφαρμογή της συνθήκης Λισαβόνας είναι κέρια σημασία το άρθρο 9 και συμφωνώ με την ανάλυση σας ότι δεν έχουμε αξιοποιήσει πλήρως μέχρι στιγμής το δυναμικό ε, του άρθρου αυτού. πέραν αυτού ε, είναι απολύτως απαραίτητο εδώ όπως και στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης ε, να ληφθεί υπόψη αυτό το σημείο και ο προβληματισμός μας να μην περιορίζεται στο ΕΠΣΚΟ ε, θα πρέπει να εμπνεύσουμε και τα υπόλοιπα συμβούλια γιατί όλες οι πολιτικές πρέπει να εφαρμοστούν από κοινού. Ε, προφανώς δεν έχουν καταλάβει όλοι το, κρυμμένο, ε, το κρυφό συγγνώμη, δυναμικό του άρθρου 9. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα, το άρθρο 9, ε, η ε, οριζόντια ρήτρα, προφανώς, είναι προφανές, εξυπακούεται για μένα ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως γνώμονας αξιολόγησης του συνόλου των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δούμε ποιες επιπτώσεις έχουν στην κοινωνική πολιτική, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε πραγματικά υποεκμεταλλευόμαστε το δυναμικό του άρθρου 9 όπως είπατε και εσείς το Δεκέμβρη. Το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ θα συζητήσει την έκθεση προς ε, τον Επίτροπο για τη χρήση του άρθρου 9 και για την ε, πιο συστηματική χρήση αυτού του άρθρου 9 και την επικράτηση της διαφάνειας ε, ως προς την χρήση του άρθρου αυτού. Θα ήθελα να πλαισιώσω λίγο τη συζήτηση μιλώντας για την ποιότητα της απασχόλησης. Το 2001 ήμουν υπουργό Απασχόλησης στην προηγούμενη Βελική Προεδρία και συζητήσαμε πολύ αυτό το ζήτημα της ποιότητας απασχόλησης γιατί στο τρίγωνο της συνθήκης της Λισαβόνας ε, είχαμε την ποιότητα πάλι στην καρδιά της ε, πολιτικής απασχόλησης. Ε, χάσαμε λίγο από την δυναμική που είχαμε αποκτήσει εκείνη την ε, περίοδο. Θα μπορούσαμε να ονειρευτούμε ε, να ε, τροποποιηθεί η κατάσταση στην πολιτική απασχόληση. Στην Ευρώπη και έτσι πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι πρέπει να εργαστούμε για την ποιότητα όσον αφορά τις νέες οδηγίες, αλλά ακριβώς και της κοινωνικής προστασίας ε, που έχει και τη σημασία της. Και είμαι, έχω ακράδαντα την πεποίθηση ότι πρέπει πολλά να γίνουν για να καταστεί σαφέ ότι η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι μόνο ένα πλαίσιο για την καταπολέμηση της φτώχειας, δεν είναι μόνο ένα πλαίσιο για την προστασία των πιο απροστάτευτων, αλλά η κοινωνική προστασία είναι μια κοινωνική ασφάλιση και ένα εγχείρημα άσκηση τη αλληλεγγύη, τη αρχής τη αλληλεγγύη. Υπάρχει με διαφορετικό πλαίσιο, με διαφορετική αξία και μέτρο στα εθνικά πλαίσια, αλλά έχει πρόσθετη αξία και πρέπει έτσι να εργαστούμε και πρέπει να βασιζόμαστε σε μια τέτοια ευρωπαϊκή πολιτική. Θα έχουμε μια συνδιάσκεψη τον ε, Σεπτέμβριο του 2010 για την κοινωνική προστασία. Γιατί πώς θα, για το θα πρέπει να ερμηνευτεί η κοινωνική προστασία σε ένα αλληλέγγυο σύστημα, σε ένα σύστημα αλληλεγγύης και ένα σύστημα ασφαλήσεων και πώς μπορεί να συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση θετικά υπέρ αυτού του στόχου. Αυτό θα γίνει το Σεπτέμβριο. Θα έχουμε και μια συνδιάσκεψη για τις συντάξεις και ε, τα συνταξιδοτικά συστήματα, διήμερη συνδιάσκεψη. Και σα το λέω εξ ε, των συναδέλφων είσαστε προσκεκλημένοι. Εσεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελπίζουμε ότι θα συμμετάσχετε ενεργά σε αυτή τη συνδιάσκεψη. Διότι θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και για εσά αυτό το εγχείρημα και για μα. Και θα αλληλοϊποστηριχθούμε. Δεύτερον, οι ε, ασφαλίσει ε, και ε, οι υπηρεσίε γενικού συμφέροντο. Ευχαριστώ που συμμετείχατε στο σεμινάριο για τι υπηρεσίε γενικού συμφέροντο. Όλοι όσοι συμμετείχαν μου είπαν ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εμπειρία. Πιστεύω ότι είναι σκόπιμο και κατάλληλο να έχουμε στη διάθεσή μας μια υπηρεσία, υπηρεσίες που δεν θα περιορίζονται μόνο σε αυτά τα οποία θα είναι οι δημόσιες αγορές και δημόσιες υπηρεσίες, αλλά που θα έχουν ένα πλαίσιο που δεν θα περιορίζεται μόνο σε σχέση με τις προθέσεις της αγοράς, αλλά θα καθορίζονται οι υπηρεσίες και πρέπει να δούμε αν θα είναι οικονομικές ή κερδοφόρες από πλευράς οικονομικής ή όχι και να δούμε πώς θα εντάσσονται στην ενιαία εσωτερική αγορά μέσα στο, από την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Εδώ έχουμε λοιπόν την Οικονομική και Κοινωνική Ένωση και πρέπει να βασιστούμε σε ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αναφέρατε το άρθρο 14 της συνθήκης και τι θα γίνει αν θα χρησιμοποιηθεί λυθεί αυτό. Είναι μείζον το ερώτημα ε, σε αυτό βασίζεται η ε, εργασία της Προεδρίας μας. Σε τεχνικό επίπεδο θα έχουμε αυτό το φόρουμ και θα εξεταστεί και στη συνέχεια το θέμα της ποιότητας. Η χάρτα ποιότητας, ας το πω έτσι, οι απαιτήσει για την ποιότητα είναι κάτι το θετικό. Θα πρέπει να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση και στη συνέχεια για το νομικό πλαίσιο. Χρειαζόμαστε ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Εγώ πιστεύω ότι θετικό θα ήταν κάτι τέτοιο να το καταφέραμε αλλά επίσης πρέπει να συνεργαστούμε ώστε τα διάφορα κείμενα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που γίνεται λόγος για τα, τις διατάξεις ε, για αυτές τις επιτυχές ε, να μπορέσουν να ενταχθούν σε ένα νομικό πλαίσιο. Εγώ θα προτιμούσα ειλικρινά την πρώτη οδό, διότι το σημαντικό είναι να σημειώσουμε πρόοδο, να προαγάγουμε τα θέματα σε σχέση με την κατάσταση όπως έχει σήμερα, για να καταφέρουμε να σχεδιάσουμε και να καταλήξουμε σε έναν ορισμό των υπηρεσιών, κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος Στη συνέχεια, ελάχιστος μισθός. Εδώ έχουμε ένα σημαντικό ζήτημα ενώπιον μας. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η Βελγική Προεδρία θεωρεί στο σύνολό τη συνολικά ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο για τους ελάχιστους μισθούς. Το εξετάσαμε αυτό την προηγούμενη εβδομάδα στην ε, άτυπη συνάντηση των ε, Υπουργών Εύσκο διότι γνωρίζουμε ότι είναι ένα στοιχείο κλειδί για την ενεργό συμμετοχή, για να μπορέσουν να προαχθούν τα θέματα και όσον αφορά την ε, απασχόληση. Εδώ κάναμε λόγο λοιπόν για το ποιες πρέπει να είναι οι προϋποθέσεις και οι όροι πρόσβασης σε αυτά τα συστήματα ελάχιστων μισθών. Πρέπει να είμαστε όμως ανοιχτοί και ειλικρινείς. Δεν μας χειροκρότησαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και δεν ήταν ομόφωνη η αποδοχή των προτάσεών μας. Όμως από την άλλη πλευρά από τις ερωτήσεις που έγιναν, που διατυπώθηκαν από αυτή την ίδια Επιτροπή, γνωρίζουμε και βλέπουμε τη μεγάλη διαφορά απόψεων που υφίσταται σε αυτά τα θέματα και στα ίδια τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη δεν έχουν οριμάσει ακόμα για να αποδεχθούν κάποια κοινά κριτήρια. Όμως υπάρχει δέσμευση να συνεχιστούν οι, αλλα... οι ε, ανταλλαγές ε, των βέλτιστων πρακτικών. Θα είναι περίπλοκη η οδός που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Θα είναι ακαθόδης και σύνθετο το θέμα. Αλλά δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια. Εσείς εργαστήκατε επ' αυτού του θέματος. Υπάρχει και ένα κείμενο το οποίο ε, είναι δεδομένο της κυρίας Φιγερέδο που το επόμενο φθινόπωρο θα υποβληθεί επίσημα. Πολύ καλά. Εμείς λοιπόν από πλευρά μας έχουμε το εξής. Η Βελγική Προεδρία θα συνεχίσει θα δώσει συνέχεια στις εργασίες στις, της Διακυβερνητικής Επιτροπής για τους ε, ελάχιστους μισθούς και ευελπιστούμε ότι στα τέλη, στο τέλος θα υπάρξουν κάποια θετικά αποτελέσματα. Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντα ότι έχουμε τις κατευθυντήριες γραμμές όπου γίνεται λόγος ακριβώς για τις, τους ελάχιστους μισθούς. Στην οδηγία υπαριθμών 10 που αφορά μια νέα κατεύθυνση για την απασχόληση έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό κείμενο. Γίνεται εδώ λόγος για την πρόσβαση για τις υγειονομικές υπηρεσίες, για ένα ελάχιστο μισθό. Γίνεται λόγος για μια προσπελασιμότητα, την πρόσβαση σε μια ολόκληρη σειρά υπηρεσιών για, ένα, για το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών. Και αυτό είναι σημαντικό. Παράδειγμα, όσον αφορά το, την παροχή φυσικού αερίου και διασφάλιση της τροφοδότησης κτλ. Πιστεύω ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα μπορούσαν να δώσουν βάση και ένασμα σε μια νέα προώθηση αυτών των θεμάτων στην Ευρώπη. Εμείς θέλουμε αυτός να είναι ο δικός χάρτης για να καταλήξουμε σε μια νέα διάσταση στην Ευρώπη και ε, χρειαζόμαστε το έργο που κάνετε εσείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η εργασία που επιτελείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εργασίες του Συμβουλίου να συγκλίνουν όσον αφορά αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, αυτή τη γραμμή της οδηγίας 10, ώστε έτσι να έχουμε ένα πλαίσιο στη διάθεσή μας. Ένα πλαίσιο το οποίο θα μας δίνει τη δυνατότητα να σημειώσουμε κάποια πρόοδο. Και κυρίως κυρίως το τονίζω, σε αυτό το θέμα το οποίο είναι τόσο περίπλοκο και ευαίσθητο όπως η ελάχιστη μισθή. Τούτων λεχθέντων, θα ήθελα να πω ότι επίσης διατυπώθηκε μια ερώτηση για τους διασυνοριακά εργαζόμενους, διαμεθοριακά εργαζόμενους, για τη δυνατότητα για τη μεταφορά των δικαιωμάτων τους, αλλά γι' αυτό θα δοθεί ο λόγος στον συνάδελφο στη συνέχεια. Θα ξεκινήσω με τη μεταφορά των δικαιωμάτων. Θα ήθελα σχετικά με αυτό να πω ότι είναι ένα θέμα που έχει ιδιαίτερη σημασία ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και τις συντάξεις. Η Επιτροπή στην Πράσινη Βίβλο έχει δίκιο, διότι πιστεύω ότι αυτό είναι ο τύπος του θέματος, ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται από πλευράς μας παρότι είναι αυτονόητο ότι έχουμε και την αρχή της επικουρικότητας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, αλλά αυτού του είδους τα θέματα δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, διότι έχουμε διασυνοριακά εργαζόμενους, αλλά επίσης έχουμε από την άλλη πλευρά και άτομα που κάθε φορά είναι όλο και πιο ε, κινητο, κινούνται περισσότερο, είναι όλο και περισσότερη η κινητικότητά τους. Για να δώσω ένα παράδειγμα, Όταν, ε, εξετάζοντας αυτό το θέμα θα ήθελα να σας πω επίσης ότι αυτή τη στιγμή έχουμε διάφορα, διαφορετικά καθεστώτα για τη συνταξιοδότηση που ισχύουν από πλευρά εθνική νομοθεσία των κρατών μελών. Ξέρετε ότι είχε μια πρόταση οδηγία του 2007 που στόχο τη ήταν να θεσπιστούν ελάχιστοι όροι και προποθέσει για την μεταφορά και τη δυνατότητα μεταφορά των δικαιωμάτων συντάξεων. Αυτό το κείμενο δεν μπόρεσε να εγκριθεί γιατί δεν υπήρξε ομοφωνία επ' αυτού στο Συμβούλιο. Θα έπρεπε λοιπόν να δοθεί μια νέα πρόθεση στο θέμα αυτό, να προαχθεί εκ νέου, ώστε να ευρεθεί βρεθεί μια λύση για τους ε, ε, διακινούμενους εργαζόμενους που διασυνοριακά εργάζονται. Και νομίζω ότι ενδιαφέρον είναι να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Συντάξεων για αυτούς τους ε, ιδιαίτερα διακινούμενους εργαζόμενους. Παράδειγμα και για κάποιους επιστήμονες ακόμα. Έχει γίνει μια μελέτη για την βιωσιμότητα ενός πανευρωπαϊκού τέτοιου ενωσιακού ευρωπαϊκού συνταξιωτικού συστήματος. Εξαιρετική μελέτη και που με αυτόν τον τρόπο μια και συντάχθηκε ήδη το 2010, έχουμε κάτι στα χέρια μας. Όλοι όσοι ενδιαφέρονται σε αυτό το θέμα μπορούν να συμβουλευτούν αυτή τη μελέτη ακριβώς και να δουν τι αναφέρει. Διότι πρέπει να σημειωθεί πρόοδος αναφέρω και πιστεύω ότι από πλευράς του Επιτρόπου έχει δίκιο ο Επίτροπος θέτοντας αυτό το θέμα μεταξύ άλλων που έθεσε. Εκείνο που θα ήθελα να πω ότι είναι ότι υπάρχουν διάφορες ε, παρεμβάσεις που έγιναν και οι οποίες αναφέρθηκαν σε ένα θέμα προβληματικό και έχω συνειδητοποιήσει ότι είναι δύσκολο, ακαθόδες αυτό το ζήτημα. Αναφερθήκατε στο μέλλον των συνταξιοδοτικών συστημάτων και των συντάξεων. Πώς θα επιλύσουμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Πάντα έλεγα και αναφερόταν ότι υπάρχει κυρίως εδώ ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα όσον αφορά την η οικονομική ανάκαμψη και τα δημόσια οικονομικά. Διότι εδώ έχουμε πώς να το πω, ένα δίλημα σε σχέση με την χρηματοδότηση, την ε, χρηματοοικονομική διακυβέρνηση ε, και για την ασφάλεια που είναι ένα θέμα μίζωνο σημασία για τις συντάξεις και σε μια κατάσταση χρηματοοικονομικής κρίσης πάλι επίσης είναι σαφές και εδώ έχουμε τη συνάδελφο που ασχολείται με αυτά τα θέματα, έχουμε την συνολική διακυβέρνηση δεδομένης μιας ιδιαίτερα αρνητικής συγκυρίας σήμερα και κάθε φορά όλο και περισσότερο θα πρέπει πρέπει να το συνειδητοποιούμε αυτό. Κάθε φορά που καταφέρνουμε ένα άνεργο να εργάζεται, να βρει θέση εργασία, αυτό σημαίνει 18.000 ευρώ επιβάρυνσης για ένα άτομο ετήσια. Φανταστείτε τώρα εδώ σε αυτή την οικονομική κρίση με εκατομμύρια ανέργου τι συμβαίνει, τι κονδύλια χρειάζονται για την κοινωνική ασφάλεια, ασφάλιση και θα ήθελα να ζητήσω 20 δις ευθύς εξ αρχής για την χρηματοδότηση των συντάξεων σε μια χώρα τόσο μικρή σαν το Βέλγιο για να φανταστείτε την εμβέλεια, την διάσταση αυτού του προβλήματος. Το αναφέρω αυτό επειδή όλα αυτά έχουν επιπτώσεις άμεσα στα δημοσιονομικά, στον προϋπολογισμό. Έτσι μεταξύ άλλων πρέπει πρώτα απ' όλα αυτή τη σκέψη να κάνουμε και αυτή την παράμετρο να διασφαλίσουμε. Και πιο πέρα στη συνέχεια σε σχέση με το Βέλγιο έχουμε ε, μέχρι την τα 75 χρόνια ε, δυνατότητα να εργάζονται οι εργαζόμενοι. Αλλά η πραγματικότητα είναι στα 60, πολλοί αποχωρούν και συνταξιοδοτούνται. Και αυτό πάλι συνεπάγεται ένα μείζον πρόβλημα για μας. Τι θα κάνουμε λοιπόν εμείς. Εμείς είμαστε υπέρ της αρχής ότι πρέπει να διασφαλιστεί, με συγχωρείτε, όχι 75 αλλά 65 ετών η ηλικία συνταξιοδότησης. Και θα θέλαμε να πετύχουμε να μην ε, συνταξιοδοτούνται ακριβώ ακριβώς τα 65 χρόνια οι εργαζόμενοι αλλά να παραμένουν λίγο παραπάνω από τα 65 χρόνια στην ενεργό εργασία. Και έχουμε και την έκθεση για την υπεργύρανση που λέει ότι θα πρέπει 2 ή 3 χρόνια πέρα από αυτό το όριο των 65 ετών να μπορούν να εργάζονται οι ε, εργαζόμενοι. Αυτό μας δείχνει το θέμα πώς έχει και πώς θα καταφέρουμε να το πετύχουμε. Αυτό είναι το ερώτημα. Πώς θα καταφέρουμε να πετύχουμε αυτό τον στόχο. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε κίνητρα από πλευράς μας. Εδώ πρέπει να το δούμε. Είναι σαφές ότι όλα εξαρτώνται, έτσι δεν είναι, από το πώς συνειδητοποιεί κανεί τα πράγματα. Αν κάποιο συνταξιοδοτηθεί στα 60 παίρνει ένα χ ποσό, στα 61 χ συν 1, στα 62 χ συν 2. Η επιτυχία τέτοιου ε, είδους μέτρων που πρέπει να είναι ε, δημιουργικά είναι σαφής. Με, αν έχουμε επιτυχία με τέτοιου είδους κίνητρα, ε, τότε λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ίσως τα καταφέρουμε. Αν δεν έχουμε επιτυχία θα πρέπει να αναθεωρηθεί αυτή η στρατηγική και θα πρέπει να σκεφτούμε κάποια συστήματα όπως την πρόορη συνταξιοδότηση. Γιατί εδώ και πάλι έχουμε άτομα τα οποία για παράδειγμα εγκαταλείπουν την εργασία τους, τον, κόσμο, τον χώρο της εργασίας στα 50 χρόνια. Με την πρόορη αυτή ε, συνταξιοδότηση, αν τα άτομα αυτά φύγουν ε, με ηλικία 50 ετών και δούμε ότι αν υπάρχουν κίνητρα τα οποία θα προσφέρονται μόνο αν κάποιος ε, περιμένει ως τα 60, 61, 62 χρόνια, ε, τότε υπάρχει διαφορά και πρέπει να δούμε τι θα πρέπει να γίνει όσον αφορά την ε, συνταξιοδότηση. Τέτοιου είδους μέτρα όταν οι εταιρείε, ε, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα ίσως μπορούν να είναι υποφελή Αλλά εδώ έχουμε ένα μείζον πρόβλημα και πρέπει να εξετάσουμε και να δούμε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί Πώς γίνεται να έχουμε τις ίδιες εισφορές ε, με το γυράσκον πληθυσμό της Ευρώπης. Όλοι έχουν επίγνωση του προβλήματος και πρέπει να βρούμε μια λύση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα ήθελα, λέει ο κύριος Δελιζέ, να ευχαριστήσω όλους τους ε, ομιλητές. Νομίζω ότι υπάρχει συνένεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υποστηρίξει τις ε, προτεραιότητες ε, της Βελγικής Προεδρίας. Υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές απόψεων, αλλά σε σχέση με τους στόχους για τα άτομα με αναπηρίες ή για τα ε, άτομα με επισφαλείς όρους διαβίωσης υπάρχει συνένεση και χρειάζεται συνεργασία για την επίτευξη των στόχων. Για τα άτομα με αναπηρίες, η επικύρωση της σύμβασης του ΟΗΕ πρώτα απ' όλα είναι σημαντική θα ασκήσουμε πίεση στα κράτη-μέλη. Με ρωτήσατε, μα δεν είναι αυτός ο στόχος απαραίτητα να ασκήσουμε πίεση στα κράτη-μέλη. Η σύμβαση είναι ε, γιγαντιαίο άλμα, είναι μια ε, σημαντικότατη πρόοδος ε, που απηχεί την άποψη των πολιτών της ε, ευρωπαϊκής κοινωνίας. Ε, τον Νοέμβριο θα γίνει ανταλλαγή των βελτίστων πρακτικών ε, και θα προσπαθήσουμε όλοι να πιέσουμε για να επικυρώσουν τα κράτη-μέλη τη σύμβαση και είναι το εφαλτήριο, δεν είναι ο ίστατος στόχος η επικύρωση της σύμβασης. Υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν επικυρώσει τη σύμβαση και μετά λένε «Α, θα σκεφτούμε πώς ακριβώς θα υλοποιήσουμε, τις διατάξεις». Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχουν κακόβουλα κράτη-μέλη που δεν επιθυμούν την επικύρωση της σύμβασης. Ο κώδικα διοντολογία επίση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, ούτω ώστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να προχωρήσουμε, ε, να προχωρήσουμε όχι μόνο ε, ε, ως προς την επικύρωση, αλλά και την υλοποίηση τη σύμβαση. Σε πολλά επίπεδα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε. Ε, μιλήσαμε για την πρόσβαση στα λεωφορεία, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τα δημόσια κτίρια, οι δημόσιες υπηρεσίε, ο εξοπλισμό, ο αθλητισμό. όλα πρέπει να είναι προσβάσιμα ε, για όλου, και όχι μόνο τα άτομα με αναπτύξη Χρειάζεται μια νέα προσέγγιση στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης. Όλοι θα πρέπει να βάλουν το λιθαράκι του στο οικοδόμημα. Το ξέρω ότι μακρηγορώ, ζητώ συγγνώμη. Όλοι νομίζω γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει λύση πανάκια που θα λύσει όλα μας τα προβλήματα. Είπανε κάποιοι ότι χρειαζόμαστε ποσοτικοποιημένους στόχους. Μα υπάρχουν αυτοί. Ε, από, στις 17 Ιουνίου ετέθη ο στόχος της μείωση του 20% ε, ε, για τους ανέργους. Αλλά χρειαζόμαστε και εργαλεία ε, αξιολόγησης ε, και Όπω είπε και η κυρία Ένκελίνξε, ε, θα πρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα την κατάσταση, ούτω ώστε σε επίπεδο διαφόρων πολιτικών να επιδιώκουμε του ίδιου στόχου, να υπάρχει συνοχή. Τέλο πάντων, δεν θέλω να μακρηγορήσω. Η παιδική φτώχεια, πολλά μέλη τη επιτροπή σα μίλησαν για αυτό το θέμα. Στι 2 και 3 Σεπτεμβρίου στη διάσκεψη που θα γίνει στο Μάξον Φαμέν, ε, αναμένονται συστάσει για την καταπολέμηση τη παιδική φτώχεια, Θα βασιστούμε στα δικαιώματα των παιδιών αλλά και σε μια πολυσχηδή προσέγγιση γιατί ε, δεν είναι θέμα μόνο εισοδήματο, αλλά και πρόσβαση στην εκπαίδευση, ε, στην κοινωνική ασφάλιση, στην περίθαλψη, στην παιδεία και ελπίζουμε πραγματικά ότι θα καταλήξουμε τελικά συμφωνία για το ελάχιστο εισόδημα που είναι ένα από τα βασικότερα σημεία. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα, Πρόεδρος. Όχι όχι, όχι, συντομότατος και περιεκτικότατος ήσασταν, δεν μακρηγορήσατε. Θα θέλαμε να σε ευχηθούμε καλή Προεδρία. Ε, είναι μία περίοδος συναρπαστική γιατί μπορεί κάποιος να προωθήσει τις ιδέες του αλλά ταυτόχρονα συνιστά και μεγάλη πρόκληση ε, η Προεδρία ε, και πραγματικά καλή επιτυχία. Θα σας υποστηρίξουμε στις προσπάθειές σας. Συνάδελφοι, σας προτείνω αμέσως να περάσουμε στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης. Θα ε, ψηφίσουμε την έκθεση του συναδέλφου μας, ε, του κυρίου Τσάμπα Ορή, που δεν είναι εδώ ακόμη. Α, τι θα γίνει. Πού είστε κύριε Ορή. le vote de votre euh, δεν μπορούμε να αρχίσουμε την ε, ψηφοφορία για την έκθεσή σας χωρίς ε, να είστε παρόν. Ήρθατε, πολύ ωραία. Λοιπόν, κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησεις των κρατών μελών. Αυτό είναι το αντικείμενο της έκθεσής σας. Έχουμε επίσης δύο γνωμοδοτήσεις από την Επιτροπή Απασχόλησης και από την Επιτροπή Γυναικών. Ε, σας παρακαλώ ε, να σταματήσετε τις κατηδίαν συζητήσεις κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Ε, λοιπόν, συμβαστική κάπα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το άρθρο 2 έχουμε το άρθρο 2α. 134 της κυρίας Τουρίναν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 133 της κυρίας Στάινερου, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 136 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 135 της κυρίας Πλόν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται για την κατευθυντήρια γραμμή 7 έχουμε την συμβαστική L ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Παράγραφος 9 της Επιτροπής Γυναικών υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Για την κατευθυντήρια γραμμή 7 πάλι. Συμβαστική M. Για την προσθήκη μιας παραγράφου. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και φτάνουμε έτσι στην τροπολογία 142 της κυρίας Τουρίνεν. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συ, τροπολογία 146 της κυρίας Τουρίνεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία όμικρον για τη δεύτερη παράγραφο της κατευθυντηρίας γραμμής 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Φτάνουμε τώρα στην παράγραφο 10 από το, της Επιτροπής Γυναικών, ένιδη ε, προσθήκης υπέρ. Σε, σελίδα 9, έχω φτάσει σελίδα 9. η παράγραφος 10 από την Επιτροπή Γυναικών είναι η προσθήκηση υπέρ παρακαλώ κατά νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά θα κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση έχετε τις ε, κάρτες ψηφοφορίας όλοι ψήφισαν όλοι έχουν όλοι τις κάρτες καταπληκτικό Πέρας ψηφοφορίας. 20 προς 27, απερίφθη, αφέστατα. Ε, κατευθυντήρια γραμμή 8 για τον τίτλο. Ε, η τροπολογία 2.29 δεν χρειάζεται να ψηφιστεί. Επανερχόμαστε στην κατευθυντήρια γραμμή 7. Δεν ξέρω για ποιο λόγο λέει η Πρόεδρος. Ε, εκα, τροπολογία 183 υπέρ κατά 183 λέω υπέρ κατά αποχές ε, σαφέστατα εγκρίνεται η 185 αποσύρεται συμβαστική π για την παράγραφο 3 της κατευθυντήριας 7 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Και τώρα ε, η 201 ήρθε, 203 της κυρίας Στάινρουκ και Γκούνς, ε, ε, ε, υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. 204 της κυρίας Στάινρουκ, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 12 της νομοδότησης Επιτροπής Γυναικών, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Nous en venons. Q. Ε, συμβαστική Q. Non, il nous faut voter. Pardon. Όχι ζητώ συγγνώμη, τη 214 της κυρίας Τουρίνεν πρέπει να την ψηφίσουμε υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τώρα... L'amendement 215, puisque l'amendement 215, γιατί η 17 αποσύρθη, υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίψετε. 216 υπέρ. Κατά. Αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. Παλήθευση για τη 216. 216. Ψηφίστε παρακαλώ. Tout le monde a Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 27 προς 22 εγκρίνεται. Η 217 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.18 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για την κατευθυντήρια γραμμή 8 έχουμε τη συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην παράγραφο 2 της κατευθυντήριας 8 στη συμβαστική Αρ, υπέρ κατά αποχές Καλά, συγγνώμη, έκανα λάθος, ευχαριστώ που είστε τόσο προσεκτικοί. Ε, υπάρχει μια προσθήκη, η παράγραψη 25 της ΕΚΟΝ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα φτάσαμε στη συμβαστική άρη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, μετά την παράγραφο 2 της κατευθυντήριας 8 φτάνουμε στην τροπολογία 248 της κυρίας Τάινρο και του κυρίου Κρίστενσεν. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 21 καταπίπτει, 242-245 έχουν αποσυρθεί. Καταπίπτουν οι λοιπές τροπολογίες γιατί καλύπτουν τη συμβαστική. 251, κυρία Τιουρίνιν και άλλων, υπέρ. Κατά Νομίζω ότι απορρίπτεται επαλήθευση, παρακαλώ. 251. Για τη 251. Ψηφίσατε. 21 ψήφι προς 28, όντως απορρίπτεται. 252 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Η 253 του κυρίου Σέρκας υπέρ. Είναι συμβατή η τροπολογία, έτσι δεν είναι κύριε Σιγητά. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 254 με τους ίδιους όρους, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 218 euh, Η 218 εγκρίθηκε. 24 καταπίπτει και η 265 και η 266 και 67 και 28 της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Πάμε στη 268 του κυρίου Ωρί. Ε, υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές θα γίνει επαλήθευση. Εδώ πρέπει να το εξακριβώσουμε. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Για τη 268 του εισηγείται. παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας. 23 ψήφι προς 26 όντως απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 269 ε, της ε, κυρίας ε, Στάινερου και άλλων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 270 του εισηγητή υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ο, ναι, εντάξει, επαλήθευση. Γιατί 270, επαλήθευση. Tout le a pu Πέρας, 25 προς 21, δίκιο είχατε. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Le 25 a été retiré. Nous votons donc le compromis S. Πάμε τώρα στη συμβαστική S υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Α. L'amendement 271 de M. Thomas θα ψηφιστεί μη προσθήκης. Είναι στη μέση της σελίδας 20 κανονικά. Μάνι, έχουμε δύο τόμες επιφανείς, έτσι, από τη Γερμανία. Ευρύτατος ο συνασπισμός. Έχουμε και τον Τόμας Χάντελ. Και το, την κυρία Τσίμερ και τον κύριο Νταγιαρέικ για τη 271. Μα είναι κατά ο εισηγητής όμως να το τονίσω. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Nous votons donc le paragraphe 29. Ε, η παράγραφος 29 της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων τώρα, υπέρ παρακαλώ. Κατά είχε συγκρίνεται. Εντάξει, να ας το εξακριβώσουμε. Παλήθευση για την ε, ε παράγραφο 29 της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι πέρας ψηφοφορίας. Καλά, άντε θα είμαι καλή αυτή τη φορά. Ας ξαναψηφίσουμε αφού δεν προλάβατε. Tout le monde est d'accord sur le vote Et tout le monde a pu voter Συγγνώμη, οι συντονιστέ ασχολούνται με το να καθοδηγήσουν την ψηφοφορία, να δώσουν τι ενδείξει. Ε, κάποιοι έχουν ακόμη ενδιασμού. Ψήφισαν επιτέλου όλοι. Αχ, εγώ δεν ψήφισα τώρα. Ξέχασα εγώ. εντάξει, τώρα νομίζω ψήφισαν όλοι. 26 ε, προς 22. Εγκρίνεται όντως. Παράγραφος 20 της Επιτροπής Γυναικών. Ε, προσθήκη, έτσι, υπέρ. Κατά απόχε. απορρίπτεται. Τίτα τι. Κυρία Τρούμπ, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Nous 293. Τώρα, 293, ε, κυρία Τουρίνεν, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 294 της κυρίας Τουρίνεν, πάλι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Εκτιμώντας ένα τροπολογία 28 του κυρίου Τόμας Χέντελ. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά το εκτιμώντα 1 έχουμε ε, την παράγραφο 1 της Επιτροπής Γυναικών υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, ε, συμβαστική α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 31 ε, της κυρία Στάινρου και άλλων υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. παράγραφος 2 της Επιτροπής Γυναικών. Υπέρ παρακαλώ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ε, παράγραφος 3 της Επιτροπής Γυναικών μετά το εκτιμώντας 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, εκτιμώντας 4 τροπολογία 33 του κ. Τόμας Χέντελ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 34 της κυρίας Φιγκρέιντο υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 35 ε, της κυρίας Δράπτη ε, και της κυρία Στάινρουκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, συμβαστική β για το εκτιμώντας 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα μετά το εκτιμώντας 5 τροπολογία 40 ε, υπέρ κατά από Νομίζω ότι απορρίπτεται η ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 40, σελίδα 22 του κυρίου Κάμπρνοχ. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι πέρας. 31 προς 14, ε, σαφέστατα εγκρίνεται. Ε, συμβαστική C. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 Madame Τώρα, τροπολογία 43, υπέρ. Κατά. Ε, θα ότι την ψηφοφορία. 43, υπέρ, υπέρ. Για 43. Κατά τώρα. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. Ε, εκτιμώντας 7, συμβαστική D, υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4 της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Εκτιμώντας 8, συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην παράγραφο 4 της Επιτροπής Γυναικών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μετά το εκτιμώντος 8 έχουμε τη συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το εκτιμώντος 8, τροπολογία 69, υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 6 της Επιτροπής ΕΚΟΝ είναι συμβατή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασ... Ε, 6 της Επιτροπής Γυναικών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά το εκτιμώντας νέα τροπολογία 77 του κυρίου Κάμπνοχ, υπέρ, κατά, αποχές, ε, επαλήθευση για την 77. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. 27 ψήφι προς 21, οπότε εγκρίνεται και πάμε στην 78 του ιδίου συντάκτη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, ε εκτιμώντας 10. Συμβαστική H υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, εκτιμώντας 11. Συμβαστική I. Ο εισηγητής μας. Παρακαλώ. Δεν υπάρχει διερμηνία δυστυχώς. Ένα λεπτό, έψαχνα το κείμενο, λέει στο κείμενο fights against, μετά το against, Μάλλον μετά το fights πρέπει να προσθεθεί το against. Against segmentation. Λείπει το against. Πρέπει να καταπολεμήσει τον κατακαιρματισμό. Το against θα προσθέσουμε. Αν συμφωνείτε θα είναι σαφέστερο το κείμενο. Οι φιλελεύθεροι, συναδελφοί μας οι φιλελεύθεροι ζήτησαν αυτή την γλωσσική προσθήκη. Σε ποιο κομμάτι λέει η Πρόεδρος. Στο τελευταίο κομμάτι της συμβαστικής, στην ένατη γραμμή από το τέλος, αυξάνει την ποιότητα, την ισότητα των φύλων, ε, καταπολεμώντας τον κατακαιρματισμό fighting against segmentation, έτσι προπαρέχοντας ασφάλεια στους εργαζομένους. Ε, είναι ούτε γλωσσική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η τροπολογία, τόσο είναι διατύπωση βελτιώνεται, δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Συμβαστική ΑΗ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα, ε, τροπολογία 100 της κυρίας Τιουρίνου και κύριου Κορνέλησεν ε, είναι προσθήκη, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 7 της ε, τη Επιτροπή Γυναικών Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά το εκτιμώντας 11, συμβαστική ΥΓΙΟΥ ε, υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, εκτιμώντας D, ε, τροπολογία 106 για διαγραφή παραγράφου υπέρ πα, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 107 της κυρίας Όμινε Ρόιτεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 108 του κυρίου Πουπάκη είναι συμβατή μου λένε, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, παράγραφος 12 από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων συμβατή υπέρ, κατά... Γιατί δεν ψηφίζετε, σταματήστε να ψηφίζετε. Υπέρ παρακαλώ, για το 12, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 110 απεσύρθη ε, για το εκτιμώντας 13 συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Παράγραφος 14 της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Αφού λέει ότι καταπίπτει, λέει ο Πρόεδρος, εφόσον ε, εγκρίθηκε η 114. Bon, allez, on va voter le 14 de la Commission économique et monétaire. Λοιπόν, τη 14 έκον, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το εκτιμώντας 13 συμβαστική τι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και μετά το εκτιμώντας 13 τοπολογία 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 115 είναι συμβατή υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το κοιμός 13, η τροπολογία 117, τη και Κορνέλισεν υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, 14, τροπολογία 120, Τόμας ε, Μαν, ε, κύριος Λέγια Ρίκ. Μα δεν είναι το κύριο Τόμας Μαν, είναι το κύριο Τόμας Χέντελ. Πω, πω, τα μπλέξα. Χάθηκα τώρα. Χέντελ, Τόμας Χέντελ. Ενσούλτιγκουν και Γερμανιστή πρόεδρο. Με το συμπάθειο. Με το συμπάθειο. Κατά. αποχέ. Απορρίπτεται. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. Μετά το εκτιμώντα 14, η 123 τη κυρία Μπλίνκεβίτσιουτε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, εκτιμώντας 15 ή 124 του κυρίου Πουπάκη Περ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 125 Τόμας Χέντελ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκτιμώντας 16 ή 127 της κυρίας Κώστα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 129 του κυρίου Χέντελ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 128 του κύριου Πουπάκη υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται ε, εκτιμώντας 17 ή 19 της έκον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά το εκτιμώντας 17 η τροπολογία 130 του κύριου Χέντελ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τώρα φτάσαμε στο τέλος της ψηφοφορίας. Θα ε, ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για το σύνολο του σχεδίου έκθεσης. Ψηφίστε παρακαλώ. Tout le monde Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Ε, Κάποιο δεν ψήφισε, αλλά μπορεί να μην θέλει να ψηφίσει. Πέρα ψηφοφορία. 40 ψήφοι υπέρ, 2 κατά 7 αποχέ. Τώρα θα ψηφίσουμε με του ίδιου όρου το σχέδιο του νομοθετικού ψήφισματο. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Tout le monde a Ψήφισαν όλοι. Τσαμπά, don't you want to vote? Le vote est clos. Πέρας. 40 υπέρ, 2 κατά. Τα ίδια αποτελέσματα. Συγχαρητήρια στον εισηγητή μας. Nous en venons au vote du rapport d'initiative de Τώρα πάμε στο σχέδιο έκθεση πρωτοβουλία τη κυρία Ρέντερ για την ανάπτυξη του δυναμικού απασχόλησης για τη νέα βιώσιμη οικονομία. Έχουμε πέντε διαφορετικές εγγνωμοδοτήσεις από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων περιβάλλοντο, Γυναικών, ε, Ήτρε Βιομηχανία και ε, Περιφερειακής Πολιτικής πριν ε, ε, την παράγραφο 1, 22 ε, της κυρίας Ζησάγια, υπέρ, κατά, άποχες απορρίπτεται. Πριν την παράγραφο 1, η 3 της Επιτροπής Περιβάλλοντος, υπέρ, κατά, άποχες απορρίπτεται. Η 1 της ίδιας Επιτροπής υπέρ Καλά, θα το επαληθεύσουμε. Λοιπόν, ξαναψηφίζουμε για την ε, τρίτη παράγραφο της νομοδότησης Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 26 ψήφοι υπέρ, 22 κατά. Εγκρίνεται, δίκιο είχατε. Λοιπόν, η ένα της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται σαφέστατα η 11 της Ρέτζη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 2 της ΕΚΟΝ. Καλά, θα ευαληθεύσουμε και την 11. Ψηφίστε παρακαλώ. Tout Πέρας ψηφοφορία. 27 pour, 20 υπέρ, 20 κατά, σαφέστατα εγκρίνεται. Ε, ε, οι δύο της Επιτροπής έχουν καταπίπτει και πάμε τώρα στην παράγραφο 1, τη συμβαστική D. Ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, τώρα, η 11 Τσέμβη, παρακαλώ, κατά αποχές απορρίπτεται, η 1 της έκον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 21 της έμβη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 1 της ήτρε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 33 του κυρίου Τόμας Μαν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 11 της ΕΚΟΝ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, παράγραφος 2 συμβαστική ε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται η, μετά την παράγραφο 2 η συμβαστική ΒΒ υπέρ. Κατά θα επαληθεύσουμε. Tout le monde a pu voter. Ψήφισαν όλοι. Le Πέρας. 20 pour, 26 contre. Ε, υπέρ 26 κατά. Μάλλον δεν είναι και πολύ συμβιβαστική αυτή η τροπολογία γιατί απερίφθη. Ε, παράγραφος 2, ε, τροπολογία 25. Παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Δεν γίνεται να έχει καταπέσει αν δεν έχουμε γκριν την προηγούμενη. Λοιπόν, 25. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, η συμβαστική έφυγε την παράγραφο 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 3, το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 6 της εκνομοδότησης Επιτροπής Περιβάλλοντος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μετά την παραγράφο 3 η 21 της Ήτρε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η 8 της Έμβη. Υπέρ. Κατά. Αποχές επαλήθευση. Επαλήθευση για την ε, παράγραφο 8 της γνωμοδότησης Επιτροπής Περιβάλλοντος. MV8. Υπέρ. Ε, ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. 21 ε, ψήφοι υπέρ, 25 κατά. Απορρίπτεται. Η 9 της ίδιας Επιτροπής υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 10 ε, της επιτροπή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 19 πάλι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εγκρίνεται, εντάξει. Συμβαστική G, υπέρ. Adopté après le paragraphe Παράγραφος 2 της ε, MV υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 4 της υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 20 της υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 5, παράγραφος 5, τροπολογία 38 της κυρίας Εσάγια υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καλά, εντάξει, επαλήθευση για 38. Le vote est ouvert sur le 38. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι πέρας. 26 υπέρ, 19 κατά, δύο αποχές. Με διαφορά εγκρίνεται. Ε, 37 Λουδίξον, 39 συγγνώμη υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 40 απεσύρθη. Τώρα θα ψηφίσουμε τη συμβαστική τροπολογία H για την ε, παράγραφο 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 6 η 14 της Ρέτζη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 6 η πρώτο τμήμα της ΕΜΒ 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 6, τροπολογία 44 του κυρίου Μάν, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 7, η συμβαστική ΑΗ, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Donc je comprends que puisque nous avons adopté le από όσο καταλαβαίνω, εφόσον εγκρίναμε τη συμβαστική ΑΕ, θα ψηφίσουμε την ΕΚΟΝ 8, αλλά θα μεταφερθεί. Δεν νομίζω υπάρχει αντίρρηση. Οπότε, ΕΚΟΝ 8, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Για την παράγραφο 8, συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση της συμβαστικής J. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Πέρας ψηφοφόρη. 26 pour, 26 υπέρ, 20 κατά, καμία αποχή, εγκρίνεται. Στο παράγραφ 8, nous en venons à au paragraphe 2 de la commission. Παράγραφος 2 της Ρέτζη, υπέρ, κατά. Ρέτζη 2, υπέρ, κατά, αποχής. Εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 21, δεν ξέρω τώρα πώς πηδήξαμε από την 8 στην 21, αλλά τέλος πάντων η τροπολογία 108 του κυρίου Πουπάκη με μια προφορική τροπολογία ούτως ώστε να μπούμε within the existing paragraph. Ε, υπέρ. Κατά αποχές η τροποποιηθήσα τροπολογία εγκρίνεται λοιπόν. Η 108 του κυρίου Πουπάκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 8 η Ρέτζι 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 12 της Ήτρε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 23 της Ήτρε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 13 Έμβη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα φτάνουμε ε, στην ε, παράγραφο 10, έκον υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, η MV7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, MV17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, η 73 της κυρίας Πλουμ υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Για την παράγραφο 9, συμβαστική και υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 9, η ήτρε 4, υπέρ, κατά, αποχές, ε, ε, επαλήθευση παρακαλώ για την ήτρε 4. Ψήφισαν όλοι. Πέρες ψηφοφορίας. 38 ψηφί υπέρ, 8 κατά, μία αποχή. Σαφέστατα εγκρίνεται. Η Ήτρε 5 μπορεί να θεωρηθεί ως προσθήκη ως προς την Ήτρε 4 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Ρέτζι 13 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 52 της κυρίας Εσάγια υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 53 της κυρίας Εσάγια υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται επαλήθευση για την 53 παρακαλώ. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 26 υπέρ, 20 κατά, εγκρίνεται. Ε, λοιπόν, έχουμε μια προφορική τροπολογία του, της εισηγήτριας για νέο τίτλο Job Potential for Women and Men in the New Sustainable Economy Δυναμικό για τις γυναίκες και τους άντρες σε μια βιώσιμη οικονομία Υπέρ παρακαλώ για την προφορική τροπολογία κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται. Tout le monde a Πέρας. 25 υπέρ, 21 ψήφοι κατά. Εγκρίνεται. Ε, να πω σε όσους ε, την καταψήφισαν, ε, αρκεί να αντιταχθείτε στην προφορική τροπολογία, ούτως ώστε να μην υποβληθεί καν σε ψηφοφορία. Παράγραφος 1, υπέρ. Της Επιτροπής Γυναικών εννοούσα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Φάμα Α, συμβατή. Άρα, ε, σαν προσθήκη θα την ψηφίσουμε. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Η ΦΑΜ 4. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Ε, για την παράγραφο 10, συμβαστική L. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 10, στην ΦΑΜ 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ΦΑΜ 19 υπέρ κατά αποχές ε, ε απορρίπτεται. ΦΑΜ 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ΦΑΜ 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΦΑΜ 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΦΑΜ 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 της ίδιας επιτροπής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 113 του κυρίου Λούντβικσον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για τον τίτλο δεν καταπίπτει αυτή όχι 64 της κυρίας Εσάγια, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, εντάξει, επαλήθευση για την 64 της κυρίας Εσάγια. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Ωραία, πέρασε. 23 ε, υπέρ, 24 κατά. Ε, Απορρίφτεται. Η για την παράγραφο 11 συμβαστική ΕΜ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, παράγραφος 12. Συμβαστική εν υπέρ. Κατά άποχες εγκρίνεται. Και φτάνουμε ε, μετά την παράγραφο 12 στην Ήτρε 24 υπέρ. Κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 12, συμβαστική όμικρον υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφο 13, τροπολογία 77 για τη διαγραφή υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 78 του κυρίου Στέρξ υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 14, σημαστική π, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, παράγραφος 15, σημαστική Q, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και μετά την παράγραφο 27 φτάνουμε στην 136 του κυρίου Πουπάκη. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 16. Συμβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 12 έχουμε την ε, τροπολογία 75 του κυρίου Κουπάκη. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 17. Τροπολογία 92 της κυρίας Κρετή υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Μετά την τροπολογία 17, τροπολογία 93 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Εντάξει, επαλήθευση για την 93. Αλλά δεν πολυψηφίζεται, δεν σας βλέπω να πολυψηφίζετε. 93. Ψήφισαν όλοι πέρας. 27 ψήφοι υπέρ, 20 κατά. Όντως εγκρίνεται. Ε, S υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μετά την ε, παράγραφο 3... Παράγραφος, ε, τροπολογία 35, συγγνώμη, του κ. Πουπάκη, με μια προφορική τροπολογία ε, προσθέτουμε το to devise in cooperation with. Σε συνεργασία με, λοιπόν, 35 συν προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η Ήτρε 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, στην παράγραφο 18 έχουμε δύο τροπολογίες για διαγραφή που έχουν αποσυρθεί, οπότε πάμε στη συμβαστική τι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, ε, συμβαστική γιου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Μετά την παράγραφο 19 έχουμε την έκον 3 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, η παράγραφος 20. Η, η συμβαστική Β υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, παράγραφος 21. Η συμβαστική W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 22 συμβαστική X υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, παράγραφος 8 της Ρέτζη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, δεύτερο τμήμα της Ρέτζη 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζη ε, 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 34 του κ. Πουπάκη υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Η 34. υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Συμβασ... Ε, παραγράφος 23 συμβαστική Y υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. φτάνουμε στην ε, τροπολογία 117 των κυρίων Εντελή και Σρέντερ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 119 της κυρίας ε, Κρετού. Ε, ως προσθήκη θα την ψηφίσουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 24. Τροπολογία 120 της κυρίας Εσάια υπέρ κατά αποχές επαλήθευση. Επαλήθευση για την 120 κυρία Σεσαΐα. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. 26 υπέρ 21 κατά. Σαφέστατα εγκρίνεται. Η 121 του κυρίου Πουπάκη υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται η παράγραφος 25 συμβαστική Z υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά την παράγραφο 25 η τροπολογία 124 της κυρίας Γκρινού και του κυρίου Πουπάκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 του κυρίου Πουπάκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έμβη 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, συμβαστική ΑΑ για την παράγραφο 26 υπέρ τα αποχές εγκρίνεται. Τώρα θα πάμε στην 135 του κύριου Πουπάκη. Με προφορική τροπολογία, αντί για green λέμε sustainable πλέον, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά, MV22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, πάμε τώρα στις παραθέσεις. Μετά το 2, τροπολογία 1 της κυρίας Σρέντερ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 2, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι 2 της εισηγήτριας, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 της κυρίας Εσάια που είναι για τη διαγραφή του 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 4 της Εσάια υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 5 της ίδιας συντάκτρες υπέρ Μάλιστα, επαλήθευση για την 4. Ε, 4 τροπολογία 4 της κυρίας Εσάγια, παρακαλώ. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 25 pour, 22. 25 υπέρ, 22 κατά. Εγώ κάνω λάθος για τα Τόμας, Τόμας Χάντελ, Τόμας Μάν και εσείς ε, και ε, κάνει λάθος όμως και το μηχάνημα. Ε, ή πατάτε λάθος κουμπί. Δύο φορές έχετε κάνει λάθος ήδη σήμερα. Μην σας γίνει και συνήθιο. Ε, όχι, δεν θα κάνουμε επαλήθευση και για την τρία, Ήταν σαφέστατα τα πράγματα. Μόνο για την τέσσερα, της κυρίας Εσάγιο. Παρακαλώ. τέσσερα. Ε, τώρα δεν θα τα ξαναψηφίσουμε όλα. Τέσσερα. Παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι πέρας. 26 υπέρ, 21 κατά, τα εγκρίνετε Η 5 της κυρίας Εσάγια υπέρ. Τι έγινε τώρα, κυρία Εσάγια Την τρία μπορούμε να την ελέγξουμε, σας παρακαλώ. Μα Κοιτάξτε, όχι τώρα είναι αργά. Δύο φορέ έχω κάνει επαλήθευση, λέει η Πρόεδρο, θα το δούμε στην Ολομέλεια. Μα ζήτησε επαλήθευση η Πρόεδρε και δεν με είδατε. Μα δεν ζητήσατε. Όχι, τελείωσε. Η έξι της Πέντε υπέρ. Κατά. Καλά, επαλήθευση. Tout Ψηφίσατε όλοι πέρα τη 26 υπέρ. 26 υπέρ 21 εναντίον εγκρίθηκε. Τώρα για την επόμενη της κυρίας Εσαγιά υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε με το ίδιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, Παύλα 1 της Επιτροπής Ήτρα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 3 ίδιας Επιτροπής υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 7 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε λοιπόν περνάμε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις β τροπολογία 8 της κ. Άγκρον υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε σε τροπολογία 9 εσαγιά με προφορική τροποποίηση θα αντικατασταθεί το EPPC με τη συμφωνία της Κοπενχάγης λέγεται. Αυτό, accord, συμφωνία στα αγγλικά. Εντάξει, Copenhagen Accord, εντάξει, έστω. Λοιπόν, είναι, ναι, όπως τοποποιήθηκε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Και μετά την αιτιολογική σκέψη C θα περάσουμε στην παράγραφο 4 της Επιτροπής ε, Περιφερειακών Υποθέσεων με προφορικές τροποποίησεις ε, γλωσσικού χαρακτήρα υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίθηκε. Μετά από την αιτιολογική σκέψη ΔΕΤΑ, η 10 της κυρίας Ομερόιτεν υπέρ κατά αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 10. Ρόιτερ, Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι και όλες πέρας ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 22 εναντίον. Εγκρίθηκε η τροπολογία 10. Περνάμε στην παράγραφο Β της Επιτροπής Ήτρε. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Στο, ε, στην αιτιολογική σκέψη Ι, ε, τροπολογία. Ε, θέλετε να ελέγξουμε. Πολύ καλά λοιπόν. Την D, της Ήτρε, παρακαλώ. Στην B της Ήτρε ψηφίσατε όλοι. Ψηφίζουμε την παράγραφο B, Β της Ήτρε. Εισηγείται εναντίον. Ψηφίσατε όλοι και όλες πέρας ψηφοφορίας. 26 υπέρ, 18 εναντίον, 3 αποχές. Εγκρίθηκε λοιπόν. Και τώρα η αιτιολογική σκέψη ε, η, η συμβιβαστική τροπολογία α, υπέρ, κατά απόχες εγκρίθηκε. Όχι, το αποτέλεσμα ήταν σαφέστατο. Εντάξει, αν αλλάζεται άποψη, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Ήταν όμως σαφές ότι εγκρίθηκε. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα ελέγξουμε. Λοιπόν, ψηφίσατε όλες και όλοι πέρας ψηφοφορίας. Και πάλι 28 υπέρ 19 εναντίον α, εγκρίθηκε. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε μετά την αιτιολογική σκέψη ε στην παράγραφο 10 Τη Ήτρε με προφορικές τροποποίησεις υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Η 14 αποσύρθηκε, ψηφίζουμε τώρα την συμβαστική τροπολογία B, Β, για την αιτιολογική σκέψη F, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Μετά την αιτιολογική σκέψη F έχουμε την 15, παράγραφο 15 της Οικονομικής Επιτροπής 15, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Μετά το f 16 τη εισηγήτριας, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Παράγραφος όχι. Η Β της επιτροπή Γυναικών υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Αιτιολογική σκέψη. Ε, συμβαστική Γ. Σ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Μετά την ε, αιτιολογική σκέψη G, η παράγραφος F της Επιτροπής Γυναικών υπέρ κατά η C της Επιτροπής Γυναικών υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίθηκε και αυτή. Και τώρα περνάμε στην παράγραφο τη Επιτροπή Γυναικών υπέρ κατά αποχέ εγκρίθηκε. Ε τη επιτροπή Γυναικών υπέρ κατά αποχέ εγκρίθηκε. 21 τη ε, κυρίας εγκρίθηκε. Ψηφίζουμε το σύνολο της πρόταση ψηφίσματος. Ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία, παρακαλώ. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Πέρας ψηφοφορία αποτέλεσμα 43 υπέρ, μία ψήφος εναντίον, τρεις αποχές. Συγχαρητήρια λοιπόν προς την εισηγήτρια. Συγχαρητήρια. Και έτσι περνάμε στη τελευταία ψηφοφορία για σήμερα το πρωί. Έχουμε την γνωμοδότηση του κυρίου Τόμας Χέντερ για τις ε, εργαζόμενες γυναίκες σε επισφαλή κατάσταση. Παράγραφος 1. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Μετά στη συνέχεια περνάμε στην 1α. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Κυρία Μαρτίν, παρακαλώ. Σε τμήματα ψηφοφορία για την τροπολογία 14 Λοιπόν, είναι κάποιο εναντίον ε, κατά του αιτήματο φιλελεύθερη ομάδα να γίνει σε τμήματα ψηφοφορία τη 14. Ε, τότε λοιπόν μπορείτε να υποβάλλετε την τροπολογία και θα σας πω μέχρι πού θα φτάσουμε σε σχέση με την Επιτροπή και τα κρατημέλη να σχεδιάσουν και εφαρμόσουν μέτρα για να διευκολυνθεί μια επαρκής ε, ε, εκπαίδευση και δυνατότητα κατάρτισης για τις νέες ε, γυναίκες όσον αφορά την εργασία τους. Εδώ, εκεί ζητώ να, μέχρι εκεί να φτάσουμε υπογραμμίζουμε μετά την ανάγκη οι γυναίκες μετά από την ε, ε, διακοπή της εργασίας τους για να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί να μπορέσουν να ληφθούν εκ νέου υπόψη. Η φιλελεύθερη ομάδα ζητεί λοιπόν σε τμήματα ψηφοφορία. Μετά από τις νέες γυναίκες θα είχαμε εκεί το επόμενο, την επόμενη παράγραφο σε σχέση με τη μετανάστευση. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ του πρώτου τμήματος κατά αποχές εγκρίθηκε το πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε τώρα το υπόλοιπο του κειμένου όπου λέγεται υπογραμμίστε επιπλέον κτλ. λοιπά. Λοιπόν, ότι οι γυναίκες όταν σταματούν την εργασία τους επειδή ε, γεννούν ένα παιδί να μπορέσουν να ξανασυνεχίσουν ιστερότερα την επαγγελματική τους ζωή. Ποιοι είναι υπέρ αυτού του δευτέρου τμήματος. πολύ καλά. Σε σχέση με την δική μας ε, τοποθέτηση από πλευρά της ομάδας μας θα έλεγα υπέρ. Αλλά ποιοι είναι υπέρ αυτού του δευτέρου τμήματος. Κατά. Αποχές. Αποτέλεσμα για να δούμε. Πρέπει να υπαλληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Λοιπόν, πέρας ψηφοφορίας, αποτέλεσμα 16 υπέρ. 11 εναντίον 19 αποχές. Λοιπόν, κερδίζουν οι αποχές, αλλά αυτό το δεύτερο τμήμα εγκρίνεται παρόλα αυτά, μετά από κάποια σύγχυση που δημιουργήθηκε πιο πριν. Έχουμε μια τροπολογία για διαγραφή στη συνέχεια στην παράγραφο 2 της κυρίας Γκέρλινγκ, υπέρ της τροπολογίας 15, κατά αποχές απορρίφθηκε. Και έτσι Περνάμε τώρα στη συνέχεια. Στην τροπολογία 16 υπέρ. 16. Ε, 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Στη συνέχεια, στην παράγραφο 2, τροπολογία 17, πλάμ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 της ίδιας συντάκτες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην παράγραφο 3, συμβαστική τροπολογία α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και μετά έχουμε από την ΚΟΕ έτοιμα να, να ψηφίσουμε μια προσθήκη. Λοιπόν, για να το δούμε. Η Ενωτική Αριστερά ζητεί μια προσθήκη στην τροπολογία 23 που θεωρείται ότι δεν καλύπτεται σε σχέση με τη συμβαστική τροπολογία Α από πλευρά συμφωνείτε με αυτή την ερμηνεία. Δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση. Κανεί δεν έχει κάποια αντίρρηση. Ψηφίζουμε λοιπόν την 23 τροπολογία ω προσθήκη στη συμβαστική Α. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίφθηκε. Και έτσι θα περάσουμε στην παράγραφο 3, στην τροπολογία 24, ο υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε, παράγραφος 4, τροπολογία 25, για διαγραφή υπέρ κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Τροπολογία 26, Κορνέλισεν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Μετά έχουμε την παράγραφο 4, τροπολογία 27, πλόμ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 28 της κυρίας Κορνέλισεν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 29 της κυρίας Γιώτοβα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 30 πλάμ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 31 πλάμ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Παράγραφος 6. <clears throat> Συμβαστική πρόταση Β υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 7. Έχουμε τροπολογίες διαγραφής 38-39-40 ε, από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Και μετά περνάμε στην τροπολογία 44, Thomas Mann, που έχει αποσυρθεί όμως. Έτσι περνάμε άμεσα στην ε, παράγραφο 8. Τροπολογία 45, 46, 47 είναι τα τόσιμες και είναι για διαγραφή. Ψηφίζουμε υπέρ αυτών κατά απόχες απορρίφθηκαν. Και έτσι, α, έλεγχος λέτε, εντάξει, 46, 44, 45, 46. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Πέρα ψηφοφορίας λοιπόν. Μάλιστα, 27 υπέρ, 20, 20 εναντίον, εγκρίθηκε λοιπόν. Εγκρίθηκαν αυτές οι τροπολογίες. Και έτσι τώρα μετά από την παράγραφο 8 περνάμε στην τροπολογία 49. Κασίν υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε μετά στην επόμενη 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Αιτιολογική σκέψη α. Συμβαστική γ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Έχουμε την τροπολογία 3, Κορνέλησεν υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Την συμβαστική δέλτα που υποβάλλεται από 5 ομάδες υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ναι, σε αυτό το σκεπτικό α έχουμε την τροπολογία 6 της κυρίας Ροντσούλη με προφορική τροποποίηση. Δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση σε σχέση με την προφορική τροποποίηση. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Το α συνεχίζουμε. Τροπολογία 7 της ίδιας συντάκτης υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 8 Λοιπόν, θα ελέγξουμε για την 7. Πολύ καλά. 7 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Πέρα ψηφοφορίας λοιπόν. Και αποτέλεσμα 26 υπέρ 21 εναντίον. Πολύ καλά. Ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Εγκρίθηκε. Ε, το υπόσχομαι. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι αυτονόητο, δεν είναι θέμα υποσχέσεων. Τροπολογία 8 της κυρίας ε, Γιώτοβα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε σαφώς τροπολογία 9 Γιώτοβα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 10 ίδια συντάξεις υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε και έτσι λοιπόν θα περάσουμε στην ψήφιση τώρα του συνόλου του κειμένου ψηφίζουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλες και όλοι και πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα 41 υπέρ, 6 εναντίον, καμία αποχή. Συγχαρητήρια λοιπόν κύριε Χέντερ. Ο κύριος, κύριε Τόμας Μαν, όχι ο κύριος Τόμας Χέντερ λοιπόν. και έτσι συγχαρητήρια και θα σας δούμε στις 3 το